morning. Good morning everybody. Καλημέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ. Ως συνήθως έχουμε τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Για λόγους προϋπολογισμού στο Προεδρείο αποφάσισε να ε, αναπρογραμματίσει κάποιες ε, συνεδριάσεις ε, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Τον Ιούνιο λοιπόν, Τετάρτη, στις 20 Ιουνίου, 9 η ώρα το πρωί και στις 3 το απόγευμα. Πέμπτη, 21 Ιουνίου, Πάλι πρωί και απόγευμα. 9 το πρωί και 3 το απόγευμα. Σεπτέμβριο, 19 Τετάρτη, πρωί και απόγευμα. 9 το πρωί και 3 το απόγευμα και το ίδιο για την 5η, 20 Σεπτεμβρίου. Οι συντονιστές συμφώνησαν σχετικά με αυτές ε, τις ημερομηνίες με τη γραπτή διαδικασία. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται το νέο πρόγραμμα. Και ξεκινάμε το σημείο νέα της ημερησίας διάταξης που έχει να κάνει με τις αποφάσεις σχετικά με τις περιουσιακές ε, σχέσεις μεταξύ συζύγων. Συντάκτρια είναι η συνάδελφος ε, ε, κυρία Εύελιν Κέπχαρτ. θα έχουμε κοινή συζήτηση των σημείων 9 και 10, αποφάσεις των τομέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρημένων συντρόφων. Συντάκτης είναι ο συνάδελφος ε, Μάικλ Κάσμαν. Θα εξετάσουμε λοιπόν αυτά τα δύο σχέδια γνωμοδοτήσεων και θα ορίσουμε την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Προτείνω λοιπόν Πρώτα να ακούσουμε σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων από την ε, εισηγήτρια κυρία Κέπχαρτ που θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής της και κατόπιν Αφού ακούσουμε και τον κύριο Κάσμαν θα προχωρήσουμε στη συζήτηση. Να σας ενημερώσω όμως ότι στις 7 Μαρτίου η Επιτροπή Τζούντι, η αρμόδια Επιτροπή, η Τζούρι, Ε, που είναι η ε, Επισουσία Αρμόδια Επιτροπή για τι ε, αποφάσει των τομέα περιουσιακών στοιχείων των καταχωρημένων συντρόφων, έχει υποβάλει αίτημα προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μάλλον προ τον Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα ε, σχετικά με την παραβίαση της αρχής της ισότητας απέναντι στο νόμο και της μη διάκρισης ε, σύμφωνα με, τον, ε, με τα άρθρα 20 και 21 του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η κυρία Κέπχαρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Ο Μάικλ Κάσμαν και εγώ συνεργαστήκαμε πολύ στενά και γι' αυτό χαιρόμαστε που μπορούμε να έχουμε κοινή συζήτηση των δύο αυτών ε, προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι θεωρούμε πολύ σημαντικό από την αρχή. Οι αποφάσει σχετικά με τι περιουσιακέ σχέσει μεταξύ συζύγων και αποφάσει των τομέα των περιουσιακών σχέσεων ε, των ε, καταχωρημένων συντρόφων ε, θα πρέπει να είναι ίσε. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει δύο ξεχωριστέ προτάσει. Διότι δεν μπορούμε να δεχτούμε την διάκριση που υπονοεί αυτό. Άλλωστε έχουμε τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Και στην ε, ισότητα αυτή υπονοείται ότι δεν ε, θα ε, αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τους καταχωρημένους συντρόφους από τους συζύγους. Στην Επιτροπή Ιούρη μήπως θα πρέπει να εξεταστεί αν θα πρέπει να αναπευθούν στην Επιτροπή οι δύο προτάσεις αυτές και να ζητηθεί μία πρόταση. Ε, αυτό θα το επικροτούσα ιδιαίτερα, ε, αν και αυτό σημαίνει ότι είτε εγώ είτε ο Μάικλ δεν θα είναι πια ε, η συγγητής. Αλλά νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το λύσουμε κοινή συνενέση. Το θέμα δεν είναι εδώ να τσακωθούμε μεταξύ μας, το θέμα είναι θέμα αρχής. Έτσι το βλέπουμε το θέμα και ίσως, ε, Μάικλ, θα έπρεπε να υποβάλουμε από την Επιτροπή μας ε, σχετική πρόταση ε, όπου να στηρίζουμε την Γιούρη στην διαδικασία αυτή. Ε, δεν γνωρίζουμε όμως το χρονοδιάγραμμα στην Επιτροπή Γιούρη, φαίνεται ακόμα να είναι ανοιχτό. Η πρόταση της Επιτροπής ε, στόχο έχει να ρυθμίσει θέματα διαχείρισης περιουσίας των συζύγων ε, στην καθημερινή ζωή ε, και όσον αφορά τον, το, το μοίρασμα της περιουσίας σε, σε περιπτώσεις μετά την λήξη της κοινής ζωής τους λόγω χωρισμού ή θανάτου. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά Ε, ο χωρισμός ε, και ο θάνατος ε, είναι περιπτώσεις διαφορετικές αλλά με τον χωρισμό ή την ακύρωση του γάμου θα πρέπει το δικαστήριο που έχει την αρμοδιότητα σε θέματα διαδοχής ε, να έχει την ε, δικαιοδοσία, παρότι δεν είναι σαφές ε, εάν θα έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία. Είναι πολύπλοκο το θέμα αυτό. Θέλαμε λοιπόν να απλοποιήσουμε το θέμα αυτό και να κάνουμε πιο σαφή την πρόταση. Οι τροπολογίες που υποβάλλω στην Επιτροπή επικεντρώνονται στα εξή βασικά σημεία, περιορίζονται στα εξή βασικά σημεία. Καταρχήν, την ε, υποχρέωση ενημέρωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα κατά το διαζύγιο ή το χωρισμό, το ε, δικαστήριο αποφασίζει σύμφωνα με το δίκαιο μιας χώρας και το ερώτημα είναι σύμφωνα με το δίκαιο ποιας χώρας ε, λαμβάνεται απόφαση. Εάν συμφωνούν ε, οι δύο, τα δύο μέρη δεν είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Μπορεί να επιλέξουν τη δικαιοδοσία αλλά είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίζεται ότι και τα δύο μέρη θα πρέπει να γνωρίζουν τις συνέπειες της επιλογής δικαίου και να μην λαμβάνει μόνο ο ισχυρότερος, ε, ε, από τα μέρη την ε, απόφαση. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ βασικά σημεία τα οποία θέλουμε να τονίσουμε στην πρόταση αυτή. Άλλωστε πρόκειται και για συζήτηση που είχαμε και σε προηγούμενες συζητήσεις, σε περιπτώσεις για παράδειγμα διατροφής και των περιπτώσεων διαζυγίου. Ε, ε ήμουνα και εγώ εισηγήτρια ε, όσον αφορά την επιλογή δικαίου στην περίπτωση διαζυγίου και ε, το ερώτημα είναι γιατί η ε, Κομισιόν δεν αναλαμβάνει σε όλες τις προτάσεις της την θέση αυτή του Κοινοβουλίου και γιατί πρέπει να την επαναλαμβάνουμε κάθε φορά. Αυτό καλό ότι ο, την Κομισιόν να το σκεφτεί. Στο άρθρο 5 έχουμε και την πρόταση υπαριθμών 8. Ο Μάικλ 8 ε, ο Μάικλ και εγώ είχαμε μια μικρή συζήτηση, ε, διότι ε, εμείς θέλουμε να ε, συμπεριλαμβάνονται κατά φθήνουσα σειρά τα ε, δικαστήρια. στα, ο λέει στα αγγλικά αυτό είναι αυτονόητο, στα γερμανικά όμως δεν είναι αυτονόητο. Ε, φαίνεται ότι η αγγλική γλώσσα σε τέτοιες περιπτώσεις έχει περισσότερες αποχρώσεις, το έχουμε συζητήσει αυτό επί μακρόν. θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε να είναι σαφές το σημείο αυτό. όπου επιλέγεται δίκαιο χωρίς να υπάρχει συμφωνία των δύο μερών ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, μια αυθύνουσα σειρά δικαστηρίων. Προτείναμε να υπάρχει και περαιτέρω δυνατότητα επιλογής η υπηκότητα ε, των μερών ε, ή το, στην περίπτωση ε, Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας να συμπεριλαμβάνεται ο τόπος συνήθους διαμονής να συμπεριλαμβάνεται. Να συμπεριλαμβάνεται δηλαδή η ηθαγένεια του αναγόμενου στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Ιλλανδία, η μόνιμη κατοικία του ή τη. Επίσης όσον αφορά το 16.1 γάμα, ε, θέλουμε και εδώ προσθήκη του δικαίου του κράτους στο οποίο τελέστηκε ο γάμος. Αν ε, ε, είναι να επιλέξει κανείς δίκαιο μετά τη σύναψη ενός γάμου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μπορεί να επιλογεί και το δίκαιο του κράτους το οποίο τελέστηκε ο γάμος. Ε, στην τροπολογία 12 έχουμε μία επιπλέον πρόταση. Ε, το δίκαιο του κράτους με τον οποίο οι σύζυγοι έχουν από κοινού τους στενότερους δεσμούς. Μπορεί αυτό να είναι το κράτος της μόνιμης κατοικίας ή μπορεί να είναι αλλού. Θέλουμε να αποφύγουμε όπως και να είναι την επιλογή του ευνοϊκότερου δικαστηρίου, το forum shopping δηλαδή. Ε, ωστόσο θέλουμε να επιτρέψουμε κάποιο περιθώριο επιλογής διότι ε, υπάρχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές. Μπορεί ε, άλλωστε να έχουμε γάμο εξ λόγω της εργασίας να ζει ο ένας σε ένα κράτος μέλος και άλλος σε άλλο θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα να επιλεγεί το δίκαιο του κράτους ε, με το οποίο έχουν ε, τους στενότερους δεσμούς. Ε, τη χώρα, για παράδειγμα, που γνωρίστηκαν ή που παντρεύτηκαν ή όπου έχουν κοινή κατοικία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διάφορες αυτές δυνατότητες που υπάρχουν και γι' αυτό έχουμε υποβάλει την σχετική τροπολογία. Άλλη μία πρόταση Ε, είναι το δίκαιο του κράτους της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής. Ε, νομίζω ότι και αυτή είναι αυτονόητη. Δεν ε, θα σας απαριθμίσω όλες τις τροπολογίες. Στο άρθρο 17 Όσον αφορά το, την επιλογή του δικαίου, ε, ελήψη επιλογής από ε, των συζύγων, το εφαρμοστέο δίκαιο ε, είναι και είναι πολύ σημαντικό εδώ να έχουμε μια φθήνουσα σειρά ακριβώ για να αποφύγουμε το forum shopping. Και έχουμε συμπεριλάβει επίσης ε, πιο κάτω το δίκαιο του κράτους στο οποίο τελέστηκε ο γάμος, γιατί για μένα είναι αυτονόητο αυτό. Αυτά νομίζω είναι τα πιο σημαντικά σημεία. Γενικά 25 τροπολογίες έχω υποβάλει. Ε, δεν, θα σας την παρουσιά, θα σας παρουσιάσω μία προσμία. μία. Οι συνάδελφοι μπορούν να θέσουν ερωτήσεις εάν έχουν. Κατά τα άλλα πάντως ε, είχα πολύ καλή συνεργασία με τον Μάικλ. και έχουμε ε, συντονίσει τις τροπολογίες μας ώστε εάν συμβεί αυτό που θέλει η Γιουρή να συγχωνευτούν τα δύο κείμενα ε, να μην υπάρχει ε, αντίφαση ανάμεσα στις τροπολογίες μας να μπορούν δηλαδή να συγχωνευτούν εύκολα τα δύο κείμενα μας και νομίζω ότι άλλωστε είναι στο πνεύμα της Επιτροπής να ακολουθήσουμε αυτή τη μέθοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Κέπχαρτ για την δεύτερη έκθεση να ακούσουμε τον συνάδελφο Μάικλ Κάσμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το πιο εύκολο είναι να πούμε ότι τα είπε όλα η κυρία Γκέπχαρτ. Πράγματι έχουμε συμφωνήσει σε μια κοινή προσέγγιση για να υπάρχει συνέπεια, συνεκτικότητα και σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που θεωρεί ότι αυτές είναι τροπολογίες που προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια ε, και ακρίβεια, ε, τις έχω και εγώ συμπεριλάβει στη δική μου έκθεση. Θα σας πω κάποια πράγματα, αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό κατ' εμέ είναι να ενισχύσουμε την αρχή για την οποία μίλησε και η Εύελιν. Φυσικά και καλωσορίζω τις προτάσεις της Επιτροπής για εναρμόνιση των περιουσιακών στοιχείων των καταχωρημένων συντρόπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έγκαιρες, ε, είναι απαραίτητες οι προτάσεις και νομίζω ότι το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης που στόχο έχει να δημιουργήσει ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και για να υπάρχει αυτός ο χώρος βέβαια πρέπει να μπορεί κανείς να μετακινείται, να κυκλοφορεί χωρίς ε, να χάνει τα δικαιώματά του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν των ζευγαριών, των χιλιάδων ζευγαριών οι οποίοι ασκούν το δικαίωμά τους ε, να ζουν και να εργάζονται σε χώρες που δεν είναι η, συνήθις, η χώρα στη συνήθις ε, διαμονής τους. Οι καταχωρημένοι σύντροφοι, τα δικαιώματα τους πρέπει να γίνονται σεβαστά. Είπε η Εύελιν ότι δεν χρειάζεται καν να υπάρχει διαφορετική πρόταση. Η αρχή της ισότητας απέναντι στον νόμο ε, είναι η ίδια, δεν αλλάζει, αλλά και η συνεισηγητριά μου αλλά και ο συγκεκριτή τη Επιτροπή Γιούρη συμφωνεί ότι θα έπρεπε να είχαν συγχωνευτεί αυτέ οι δύο προτάσει και θα έπρεπε πιστεύω να το πούμε αυτό. Χαιρετίζω ε, αυτό το αίτημα να γνωμοδοτήσει και ο Οργανισμό ε, των Θεμελιών Δικαιωμάτων ε, για να δει κατά πόσον ευθυγραμμίζεται με τις συνθήκες και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτή η πρόταση. Είναι πρόταση της Γιούρη και την υποστηρίζω και θα αναμένω με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Επί του περιεχομένου, όπως σας είπα, στόχος της δικής μου γνωμοδότησης είναι η νομοθεσία για τα περιουσικά στοιχεία, σχέσεις μάλλον των καταχωρημένων συντρόφων να είναι στο ίδιο επίπεδο ε, και έχουν ε, Γι' αυτό στην έκθεσή μου λάβει χώρα ίδιε αλλαγέ με αυτέ στην έκθεση τη Εύελιν. Σε ό,τι αφορά επίση το εφαρμοστέο δίκαιο, στι θεολογικέ σκέψει και στι ε, τροπολογίε από την 1 έως την 6 και στην 9. Λέω επίσης ότι θα πρέπει να ενημερωθούν από την Κομισιόν όλες ε, οι ενδιαφερόμενες ε, πλευρές γιατί πώς μπορεί κανείς να <clears throat> εφαρμόζει ένα δικαίωμα όταν δεν το γνωρίζει. Το ίδιο ισχύει και για την αρχή τη μη διακριτική μεταχείρισης για την εφαρμογή του κανονισμού. Ε, περιουσιακέ σχέσει λοιπόν των καταχωρημένων συντρόφων πρέπει να περιλαμβάνονται. Επιλογή δικαιοδοτικού οργάνου, το ίδιο να ισχύει για τους νυφευμένους και για τους καταχωρημένους συντρόφους, 13 και 15 τροπολογίες. Για τους καταχωρημένους συντρόφους θέλουμε να μπορούν να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο, στον βαθμό που μπορούν να το επιλέξουν και, όπως είπα, τα νυφευμένα ζευγάρια. Υπάρχει όμως μια πάρα πολύ σημαντική, ένας πολύ σημαντικός περιορισμός. Μπορεί να είναι το επιλεγέν δίκαιο, το δίκαιο ενός κράτους, το οποίο αναγνωρίζει το καθεστώς των καταχωρημένων συντρόφων. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιο να επιχειρήσει από το παραθυράκι, από την πίσω πόρτα, να στραφεί σε ένα κράτο μέλο που δεν αναγνωρίζει του καταχωρισμένου τρόφου να αναγνωρίσουν τους καταχωρημένους συντρόφους, την καταχωρημένη σχέση. Δυστυχώς υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε προς μια τέτοια κατεύθυνση. Υπήρχε μια δυσανάλογη διάταξη την οποία διαγράψαμε για απλή κατάργηση οποιασδήποτε διάταξη στον κανονισμό ε, κατά το δοκόν των κρατών μελών. Αυτό θα ήταν απαράδεικτο και το καταργούμε. Επίσης βελτιώνουμε την ασφάλεια δικαίου εν γέννη ε, στον κανονισμό και υπάρχουν οι σχετικές τροπολογίες 11 και 12. Εν κατακλείδη. Ουσιαστικά θα πω αυτά με τα οποία ξεκίνησα. Συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση της Evelyn Gebhardt. Έχουμε συνεργαστεί στενά οι δυο μας. Βέβαια είναι μια γνωμοδότηση για μια διαδικασία επί της οποίας Συμβουλευτικό είναι μόνο ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Ελπίζω αυτό να αλλάξει στο μέλλον. Πιστεύω πάντως ότι είναι σημαντικό εμεί στο Κοινοβούλιο να στείλουμε το σαφέστερο δυνατό μήνυμα, ότι δηλαδή η ισότητα είναι στο επίκεντρο, είναι στην καρδιά των αξιών που στηρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν στηρίξουμε την ισότητα, πώς περιμένουμε να ληφθεί υπόψη σοβαρά η αρχή αυτή από άλλους. Η διαδικασία αυτή λοιπόν είναι, όπως είπαμε, ομόφωνη έγκριση από το Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο, όπως είπα. 81 ε, δάφιο 3 είναι το άρθρο, η νομική βάση για τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχόμενο λοιπόν βέτο από Εθνικό Κοινοβούλιο είναι μια δυνατότητα, αλλά πρέπει αυτό να γίνει εντός έξι εβδομάδων από την έγκριση. Και ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Ελπίζω το Συμβούλιο να έχει τη σοφία, να έχει την ε, σοφροσύνη να δει ότι είναι απαραίτητε σε προτάσεις αυτές, έγκαιρες, επίκαιρε. Ξέρω ότι υπάρχει, υπάρχουν κάποιοι μόνιμοι εκπρόσωποι των ε, κυβερνήσεων εδώ στην αίθουσα, βλέπω κάποιους από δική μου χώρα τουλάχιστον, όσοι είναι θα έλεγα προοδευτικοί στο θέμα αυτό, νομίζω ότι έχουν ε, την υποχρέωση να προωθήσουν ε, τη θέση αυτή ώστε να κερδίσει την πλειοψηφία ή μάλλον την ομοφωνία στο Συμβούλιο. Αν παρακαλώ τώρα έχετε απορρίσει με στη διάθεσή σας εφόσον μπορώ να απαντήσω. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάσμα. Δεν ξέρω αν τα άλλα θεσμικά όργανα, Συμβούλιο ή Κομισιόν θεωρούν σκόπιμο να σχολιάσουν. Ακούσαμε τις δύο παρουσιάσεις. Θέλει η Κομισιόν το λόγο. Παρακαλώ μόνο σύντομα για να αρχίσει η συζήτηση μεταξύ των βουλευτών. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Σας θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους διεισηγητές ε, για τις εκθέσεις που μας παρουσίασαν σήμερα και για τις ε, τροπολογίες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εισηγητές γιατί καλωσορίζουν την πρόταση της Κομισιόν, λένε ότι είναι απαραίτητη, είναι έγκαιρη, Πράγματι, ε, πριν από ένα χρόνο εγκρίθηκε από την Κομισιόν το πακέτο των δύο προτάσεων και ο στόχος μας ήταν να τονίσουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι στην Κομισιόν να βελτιώσουμε, να διευκολύνουμε την καθημερινή ζωή των πολιτών, ανεξαρτήτως του κατά πόσον έχουν παντρευτεί ή αν έχουν μια καταχωρημένη σχέση. Και είμαστε ευγνώμονες ε, στις προεδρίες οι οποίες μέχρι τώρα ακολούθησαν την προσέγγιση και εξέτασαν τις δύο προτάσεις ως πακέτο και παράλληλα τη μία με την άλλη. Και οι δύο προτάσεις έχουν τον ίδιο στόχο. Δηλαδή, την παροχή σαφών κανόνων για διεθνή ζευγάρια. Κάτι το οποίο θα τους παράσχει ασφάλεια δικαίωση ό,τι αφορά τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Ιδίως όταν χωρίσει το ζευγάρι ή εάν πεθάνει ο ένας από τους δύο. Είναι ουδέτερες οι διατάξεις, δίνουν απαντήσεις σε τρία ερωτήματα. Ποιο είναι το δικαιοδοτικό, ποιο μάλλον δικαστήριο και τη δικαιοδοσία, ποιο δίκαιο είναι το εφαρμοστέο και πώς η απόφαση των δικαστήριων ή άλλων αρμόδιων αρχών των κράτων μελών μπορεί ε, να, αποφα... Ε, να εγκριθεί και να εφαρμοστεί η σχετική απόφαση από άλλα κράτη-μέλη. Με τις να στα τρία αυτά ερωτήματα θα δημιουργηθεί και αυτός ο κοινό χώρος δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Είναι αλήθεια ότι μπορεί κανείς να δώσει διαφορετικά διαφορετικές απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, εξού και η Κομισιόν επέλεξε ε, να προχωρήσει με δύο διαφορετικούς κανονισμούς. Ο γάμος είναι ένας παραδοσιακός θεσμός που υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά οι καταχωρημένοι σύντροφοι είναι μια έννοια λίγο σύγχρονη. 14 κράτη-μέλη έχουν αυτή τη δυνατότητα, παρέχουν αυτή τη δυνατότητα και μεταξύ αυτών των 14 οι ρυθμίσεις διαφέρουν. Λαμβάνοντα υπόψη λοιπόν αυτό το γεγονό, οι κανονισμοί δίνουν διαφορετικέ απαντήσει, ιδίω ό,τι αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο. Ίσως αυτό να σας ακουστεί κάπως διακριτικό, ότι δηλαδή δεν έχουν την επιλογή οι σύντροφοι για να διαλέξουν το εφαρμοστό δίκαιο. Όμως για το αντίθετο πρόκειται. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε στους συντρόφους είναι η ασφάλεια δικαίου. Να ξέρουν δηλαδή ότι άπαξ έχουν καταχωρηθεί ο ζευγάρι, υπάρχει εφαρμοστέο δίκαιο και αυτό θα εφαρμοστεί για την περίπτωσή τους. Υπάρχουν ουσιώδεις ε, διαφορές μεταξύ των δύο ειδών ένωσης, ε, νεφευμένη αφενός κατηγορημένης του Ρεφεφιντέρου. Εξού και η Κομισιόν θεωρεί ότι πιο αποτελεσματικό και πιο εύκολο σε αυτή τη φάση είναι να προωθήσουμε δύο διαφορετικούς κανονισμούς. Θα ολοκληρώσω εδώ και σας ευχαριστώ. Thank you. Now, let's open discussion. Και τώρα ξεκινάει η συζήτηση. Ο κύριος Ντεγιόγκος και ο δισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δύο εισηγητές για τις εξαιρετικές τους εκθέσεις. Πρόσφατα έλαβα απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Ευρωπή στις ερωτήσεις που είχα θέσει για τα ζητήματα των κατοχωρημένων συντρόφων σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία και πραγματικά απογοητεύτηκα πλήρως διότι ε, Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ είχε πει στο παρελθόν ότι η ελευθερία σε ελευθερία διακίνηση θα παρέχει περισσότερα δικαιώματα ειδικά στους καταχωρημένους συντρόφους και εδώ νομίζω ότι με απογοήτευσε με τις απαντήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι οι δύο αυτές ε, προτάσεις ιδιαίτερα σε ό,τι φορά τους καταχωρημένους συντρόφους πολύ σημαντικές αλλά Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση Κάσμαν ε, περιλαμβάνει κάποιες εκφράσεις ε, που δηλώνουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, περιορισμό στην διακίνηση που στις περιπτώσεις αυτές αφορά και τους καταχωρημένους συντρόφους. Τώρα, οι προτάσεις ε, βέβαια είναι εξαιρετικές. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένο που ο Κάσμαν διαγράφει το άρθρο 7 που ήταν και το σημαντικότερο πρόβλημα για την ομάδα μου. Ίσως ε, διαγράφοντας ε, την παράγραφο 18α που αναφέρεται ότι παρόμοια απόρρευση κλπ. Είναι κάτι που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Επίση, στο άρθρο 21 θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε κάποιες ε, διαφορετικές διατυπώσεις. Κατά τα άλλα έχω μία και μοναδική παρατήρηση, διότι θεωρώ ότι το, τα εκτιμώντας και στις δύο περιπτώσεις έκθεση Γκέπαρτ, ε, ε, εκτιμώντας 22α, όπου συμφωνώ ότι θα πρέπει η ερμηνεία του δικαίου να εφαρμόζεται σε ενωσιακό επίπεδο, αλλά αν υπάρξει ορισμός, αυτομάτως ε, ε, ε, γίνεται κομμάτι του της ενωσιακής νομοθεσίας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί αυτή η αναφορά, παρά μόνο να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ορισμός, κάτι το οποίο οδηγεί αυτόματα στην συμπερίληψη αυτού του ορισμού στο ενωσιακό δίκαιο. Πάντως πιστεύω ότι αυτές οι δύο εκθέσεις ε, θα πρέπει πολύ ήπια και Μαλακά να περάσουν στην αρμόδια επιτροπή. Ευχαριστώ. κυρία Ίνβελτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές. Στο παρελθόν είχα συνεργαστεί με την κυρία Γκέπχαρτ για μια άλλη πτυχή του ίδιου θέματος και πράγματι συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση της. Είναι παρόμοια ή θα έλεγα ταυτόσιμη με αυτή που είχε ακολουθήσει σε προηγούμενες εκθέσεις επί του θέματος. Θα ήθελα να ενθαρρύνω το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τις συστάσεις μας και να εγκρίνουν μια διευθέτηση του θέματος, διότι αν δεν υπάρχει ρύθμιση τότε αναλαμβάνουν τα δικαστήρια και οι μοναδικοί που υποφελούνται είναι οι δικηγόροι στην περίπτωση αυτή. Τα, θέλουμε τα ζευγάρια, οι σύντροφοι να μπορούν να υποφεληθούν Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με την πρότασή σας ε, να συγχωνευτούν οι δύο εκθέσεις σε μία και ζητάμε από την Κομισιόν να επιστρέψουμε μια νέα πρόταση η οποία θα συμπεριλαμβάνει και τις ε, δύο μέχρι τούδε προτάσεις. Η καταχωρημένη σύντροφοι όπως υπόθηκε είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο αλλά τα 14 κρατημέλη τα οποία ισχύει αυτό το σύμφωνο έχουν ε, ε, διαφορετικές νομοθεσίες και, αλλά και ο γάμος ε, διέπεται από διαφορετικά δίκαια. Και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις ε, που αφορούν στη γαμική σχέση διαφέρουν. Δεν θα πρέπει λοιπόν ο γάμο να αντιμετωπίζει με τρόπο διαφορετικό από ότι τα καταχωρημένες, τους καταχωρημένους συντρόφους. Και ελπίζω ακόμα και τελικά, πέραν από το πεδίο χαραμογής αυτού των εκθέσεων, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο και προσφάτως κιόλας, τα κράτη-μέλη που δέχονται την ε, γάμμα ανάμεσα στο άτομα του ιδίου φίλου που έχουν τον καταχωρημένη ε, καταχωρημένου συντρόφους ε, να προχωρήσουν στην αμοιβή αναγνώριση. Εντάξει, μπορούμε να δεχτούμε την αναγνώριση ας πούμε, σε ό,τι φορά την μπύρα και τα τυριά και όχι τους γάμους μεταξύ προσώπων ιδίου φίλου. Εμείς ε, λέμε ότι εορτάζουμε την ε, ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα γιατί όχι να μην ε, μπορέσουμε να γιορτάσουμε και σε αυτή την περίπτωση τους καταχωρημένους συντρόφους. Ο κύριος Γιακολίνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε δεν υπάρχει καμία εμβολία ότι οι δύο προτάσεις ε, οι οποίε είναι στενά συνδεδεμένες όπως αυτές που ακούσαμε από τους δύο εισηγητέ, θα πρέπει να προχωρήσουν ε, χέρι-χέρι και θα να έχουμε προβλέψει δύο διαφορετικές προτάσεις ε, ενδεχομένως να μπορεί να θεωρηθεί με, ως θετικό αλλά και ως αρνητικό. Δηλαδή, σας διευκρινίζω περί ομιλώ. Τώρα, το ένα αφορά το περιουσιακό καθεστώς ανάμεσα στους ε, εγγάμους, σε μια οικογένεια κλπ. Κάτι το οποίο είναι ε, προσδιορισμένο από τις νομοθεσίες. Τώρα το ζήτημα των καταχωρημένων συντρόφων είναι κάτι το καινούριο. Είναι γεγονός ότι μόνο 14 κράτη-μέλη έχουν αναγνωρίσει αυτό το καθεστώς και όχι τα υπόλοιπα αλλά προκειμένου για θέματα περιουσιακά ίσως μια ενιαία πρόταση θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί ως ε, καταλληλότερη μέθοδος για τη διευθέτηση αυτών των ζητημάτων που εμπέσχετος παραμένουν διακριτά. Τώρα σε σχέση με τον πρώτο ζήτημα οι σύζυγοι μπορούν να επιλέγουν ε, το το δίκαιο του κράτους στο οποίο κατοικούν. Υπάρχει φυσικά ε, ελευθερία εγκατάστασης. Υπάρχει και ε, το θέμα το διασυνοριακό, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, δηλαδή το 2012 μόνο το ίμιση των κρατών που να έχουν αναγνωρίσει τους, ε, τους, καταχωρημένους, τους καταχωρημένους συντρόφους, αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει σε ένα, κάποιο προβληματισμό. Διότι ο προβληματισμός υπάρχει και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Ούτε θα μπορούσαμε να παρακάμψουμε αυτόν τον προβληματισμό. Κάποιες χώρες, ε, συμπεριλαμβανομένες και της δικής μου, έχουν ε, δηλώσει ότι οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου και ε, την ε, κλασική οικογένεια. Ξέρετε ότι υπάρχει τώρα πια μια παγιωμένη θέση του, του δικαστηρίου πάνω στα ζητήματα αυτά σε ό,τι αφορά το καθεστώς που εφαρμόζεται στις ε, δραστηριότητες που μπορούν να καταγραφούν, να καταχωριστούν. Το πρόβλημα λοιπόν παραμένει και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί και να επιληθεί αλλά πώς ε, λαμβάνεις υπόψη την ε, νομοθεσία και την νομολογία που έχουμε να προβλέπουμε μια διευθέτηση συμβατική για τα ζεύγη τα οποία δεν ε, δεσμεύονται με τα, μάλλον δεν δεσμεύονται τα δεσμά του γάμου και εμβασιτώσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως ε, στην Ιταλία υπάρχουν ε, κάποιες διευθετήσεις ε, για θέματα που αφορούν την υγεία αλλά και άλλες καταστάσεις που λαμβάνουν υπόψη. Εγώ είμαι κατά κάθε μορφής διακρίσεων, κάθε μορφής και κάθε έννοιας που παραβιάζει το ζήτημα της ε, της διακριτικής μεταχείρισης. Το ζήτημα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό, πολύ λεπτό, αλλά και ευαίσθητο παράλληλα. Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μία διευθέτηση πάντως ε, των περιουσιακών σχέσεων θα πρέπει να υπάρξει και με βάση φυσικά τα όσα προτείνουν οι δύο εισηγητές, κυρία Βέμπερ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια ερώτηση σήμερα. Αλλά προηγούμενα να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές και να πω πως ε, θεωρώ και εγώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα νομοθέτημα και όχι δύο διαφορετικά. Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με τους εαυτούς μας, και θέλουμε να, να προωθήσουμε την ε, ιδιαιτερότητα και τη διαφορετικότητα Δεν θα πρέπει λοιπόν να είμαστε υποκριτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι οι διαφορές είναι σημαντικές. Σε μια χώρα υπάρχουν, ε, επιτρέπονται οι γάμοι, σε άλλη όχι, αλλά ταυτόχρονα διερωτώ πώς θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα στην χώρα μου. Στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες ε, ετέθησε εφαρμογή ο νέος ε, αστικός κώδικας και αναφέρει ότι δεν αναγνωρίζει τις ε, καταχωρημένες, τους καταχωρημένους συντρόφους Κοιτάξτε, είμαι κάπως... Ε, τα έχω τα πράγματα συγκεχημένα στο μυαλό μου, γι' αυτό και δεν μπορώ να εκφραστώ σωστά. Υπάρχουν άρθρα τα οποία είναι αντιφατικά στον ε, νέο αστικό κώδικα. Λοιπόν, εάν αυτές οι εκθέσεις εγκριθούν, τι, πώς θα, γίνει με, τις, με τα ζευγάρια τα οποία θα έχουν καταχωρηθεί ως ε, σύντροφοι σε μια ευρωπαϊκή χώρα και θα μετακινηθούν στη χώρα μου να ζήσουν. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Δεν βλέπω άλλους ευρωβουλευτές που να ζητούν το λόγο στο θέμα αυτό. Ας επανέλθουμε λοιπόν στους δύο συντάκτες μας, αν θέλουν να ολοκληρώσουν έχοντας ακούσει ε, τις παρεμβάσεις των ε, ευρωβουλευτών. Κύριε Κέπχαρτ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ε, πολύ καλή συζήτηση που είχαμε μόλις τώρα. να ευχαριστήσω και την Σοφή. Είναι σαφές, πάντα προσπαθώ στην ε, δουλειά μου να ακολουθώ την ίδια γραμμή, να μην ε, ε, προχωρώ σε αντιφάσεις. Γι' αυτό είναι σαν ντεζαβί σήμερα, διότι έχουμε ήδη συζητήσει το θέμα των διαζυγίων και το θέμα των της κοινή περιουσίας. Ε, ξέρω πόσο δύσκολα είναι τα θέματα αυτά στα κράτη-μέλη και ε, θα πρέπει να εξετάσουμε το κάθε θέμα ξεχωριστά. Προσπαθούμε όμως ε, να διατηρήσουμε κάποια συνέπεια ώστε να μην προκαλούμε σύγχυση στους πολίτες. Προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για ανθρώπους που έχουν ένα πρόβλημα επειδή παντρεύτηκαν στην περίπτωση διαζυγίου, χωρισμού ή θανάτου. Θα πρέπει να γνωρίζουν ποιο δίκαιο ισχύει και δεν ε, θα πρέπει να υπάρχουν αντιφατικές αποφάσεις και διαφορετικές αποφάσεις ε, σε διάφορα κράτη-μέλη. Αυτή την κατάσταση θέλουμε να λύσουμε και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε με τρόπο ε, μοντέρνο και σύγχρονο και προοδευτικό. Ο Μάικλ θα συμφωνήσει μαζί μου. Ε, κύριε Γιακολίνο, φροντίσαμε να ε, λάβουμε υπόψη μας την επικουρικότητα. Δεν θέλουμε να ε, επέμβουμε στο δίκαιο των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο Ευρωπαίος νομοθέτης. Αυτό που κάνουμε είναι ότι δίνουμε στον κόσμο μέσα για ε, να λύσουν τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Και στα κράτη-μέλη υπάρχουν πολύ διαφορετικές ρυθμίσεις και για ε, τον γάμο και για την ε, κοινή περιουσία. Υπάρχουν πολύ διαφορετικές διατάξεις και επίσης είναι πολύ διαφορετικό το τι ισχύει όσον αφορά τις καταχωρημένες, τους καταχωρημένους συντρόφους στα άρθρα 27 και 6 ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, περιγράφεται τι γίνεται ε, εάν ε, το δίκαιο ενός ε, κράτους μέλους είναι διαφορετικό από αυτό που επιθυμούν οι συγκεκριμένοι πολίτες. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε τον κατακερματισμό στις περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρξει κάποια συγχώνευση και ε, εκεί που υπάρχει δυνατότητα επιλογής δικαίου. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί στον ε, τομέα του δικαίου για την ε, γαμήλια περιουσία, την κοινή περιουσία. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής και όχι στην περίπτωση των καταχωρημένων συντρόφων. Ε, αν υπάρχει διαφορετικό δίκαιο όσον αφορά ε, τους καταχωρημένους συντρόφους στα διάφορα κράτη-μέλη, ε, θα πρέπει όπου υπάρχει δυνατότητα επιλογής να υπάρχει δυνατότητα αυτή, εφόσον υπάρχει και στην περίπτωση των γάμων. Το είπε ο Μάικλ αυτό ε, και πιστεύω ότι έχουμε λάβει υπόψη μας τα θέματα αυτά. Και θα ήθελα να φέρω αντίρρηση σε αυτό που είπε η Κομισιόν σχετικά με το γιατί δεν συγχωνεύει τις δύο προτάσεις. Ε, το δίκαιο που διέπει τους γάμους ενδιαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και το ίδιο ισχύει και, στις, ε, και για τους καταχωρημένους ε, συντρόφους. Αυτό λοιπόν δεν είναι ε, επιχείρημα, διότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ε, και όσον αφορά το δίκαιο που διέπει γάμου γάμους ε, στα διαφορετικά κράτη-μέλη. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό ότι διαφέρουν τα δίκαια μεταξύ τους. Το επιχείρημα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τους καταχωρημένους συντρόφους από κράτο μέλους σε κράτους μέλο δεν στέκει. Η μόνη διαφορά είναι ότι υπάρχει ο γάμος ως θεσμός και στα 27 κράτη-μέλη, ενώ δεν υπάρχουν οι καταχωρημένοι σύντροφοι ως θεσμός και στα 27 κράτη-μέλη, αλλά και αυτό το έχουμε λάβει υπόψη μας. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να το ξασκεφτούν το επιχείρημα αυτό. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που είχα. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάσμαν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Εύελιν κάλυψε τα περισσότερα από τα νομικά θέματα. Θα ήθελα να πω στους συναδέρφους ότι ο κανονισμός για ε, ε, τους καταχωρημένους συντρόφους ισχύει σε όλους τους καταχωρημένους συντρόφους. Δεν ε, αφορά μόνο τους ομόφυλους. Κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να μην παντρευτούν αλλά να έχουν καταχωρημένο σύντροφο. όπως είπε η Σοφή, το θέμα είναι να αναγνωρίσουμε ε, τα δικαιώματα και τις ευθύνες ε, σε περίπτωση που ενώνονται δύο άνθρωποι. Είναι σαν ε, μια ε, αστική ε, σύμβαση. Εγώ ως ομοφιλόφιλος θα ήθελα να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα ήθελα όταν φεύγω από την πρεσβεία μου στην Πολωνία να έχει ο σύντροφός μου τα ίδια δικαιώματα που θα έχει ένας σύζυγος όσον αφορά την περιουσία μου, την κηδεία μου, τα ε, ε, που υπάρχουν στην Πολωνία αλλά ε, το θέμα είναι ότι όταν έχουν δεσμευτεί δύο άνθρωποι να ε, βρίσκονται μαζί, ε, δεν βλέπω το λόγο να κάνει κανείς διαχωρισμό ανάμεσα στα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών που δημιουργούν έτσι τα βασικά δομικά στοιχεία της κοινωνίας. Τα δικαιώματα και οι ευθύνες που συνεπάγονται τέτοιες δεσμεύσεις πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίζονται. Κύριε ε, Βέμπερ, δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας, αλλά οι αντιφάσεις αυτές υπάρχουν και ε, στην περίπτωση του ε, δικαίου για το γάμο και στην περίπτωση των καταχωρημένων συντρόφων. Ε, όπως ε, σωστά υπόθηκε, αποτελούν ε, αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θέλω να συνεργαστώ με όλους εδώ πέρα. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να κερδίσουμε, επιφέροντας νομική βεβαιότητα και αναγνωρίζοντας τη διαφορετική προσέγγιση των διαφόρων κρατών μελών, ακολουθώντας όμως και τη δουλειά που έχει κάνει ένας πρώην συναδελφός μας, ένας Ιταλός από το ΕΛΚ, που εργάστηκε πάνω στο θέμα της οικογενειακής επανένωσης. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια προσέγγιση που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Είχε να κάνει με την επανένωση όλων ε, των οικογενειών χωρίς ε, διακρίσεις, εκτός από τις ε, διακρίσεις που υπήρχαν τότε στο δίκαιο των διαφόρων κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος να προχωρήσουμε. Dennis De Θα ξανακοιτάξω την τροπολογία για το 18.1α ως Άγγλος. Εγώ λέω ε, may not ε, δεν μπορεί, ενώ θα πρέπει να λέμε shall not, ε, θα πρέπει να λέμε ότι δεν το κάνει, δεν θα πρέπει να είναι προαιρετική η διάταξη αυτή. Πάντως είναι πολύ λεπτό το θέμα αλλά θέλω να αφαιρέσω τις διαφορές από την ισότητα και να δω αν μπορούμε να έχουμε μία ε, βασική αρχή που να καλύπτει τον γάμο και τις κατοχωρημένες ε, σχέσεις, που να ενθαρρύνει τον κόσμο να δεσμεύονται, ε, να συζήσουν χωρίς να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη να αλλάξουν το δικαιό τους. Πιστεύω ότι έχουμε τη βούληση και τη δυνατότητα να το πετύχουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο, και την κυρία Κέπχαρτ και τον κύριο Κάσμαν. Έτσι ολοκληρώνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων ε, για το σχέδιο γνωμοδότησης. ορισμός για την κατάθεση, ε, η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 11 Απριλίου 12 το μεσημέρι. 11 Απριλίου, 12 το μεσημέρι. Να θυμόμαστε ότι η ψηφοφορία στην ΛΥΜΠΕ για τα σχέδια γνωμοδότησης προβλέπεται 31 Μαΐου. Εάν όλα αυτά είναι εντάξει, προχωράμε στο επόμενο θέμα που είναι το υπαριθμόν 11 στην ημερήσια διάταξη. Έχει να κάνει με τον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότυπες διευθύνσεις σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η συγγήτρια είναι η κυρία Ρενάτε Βέμπερ. Θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων πάνω σε έκθεση πρωτοβουλίας. Μιλάμε για τις πρότυπες διευθετήσεις σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καλωσορίζουμε τον κύριο Σόιερ που εκπροσωπεί την ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου ε, του Δικαίου της Ευρώπης ε, για τα μέσα μας και στο Σαρμπρούκεν. Είδαμε ότι ένα φυλάδιο σχετικά με τη φύση και τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου αυτού έχει διανεμηθεί μεταξύ ε, έχει διανεμηθεί στους ε, συμμετέχοντες ε, στη σημερινή συνεδρίαση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το Ινστιτούτο κάνει μελέτες σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις υποχρέωσεις, τους, τα δικαιώματα των πολιτών ε, να είναι απόλυτα ενημερωμένοι. Ο κύριος ε, Σόγερ θα μας παρουσιάσει τα προσωρινά αποτελέσματα αυτής της μελέτης ε, που συνεχίζεται και επίσης έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε τον εκπρόσωπο της ομάδας υψηλού επίπεδου για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον πλουραλισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την έκθεση θα παρουσιάσει ο κύριος Γκέραρτ Ντεγκράφ από την Γενική Διεύθυνση για την Κοινωνία της ε, πληροφορίας ε, και το διαδίκτυο της Κομισιόν. Είναι διευθυντής, ε, δηλαδή αρμόδιος για το σχετικό θέμα. Θα μας παρουσιάσει μια επισκόπηση των πρώτων συναντήσεων της ομάδας υψηλού επίπεδου. Προτείνω λοιπόν να ακούσουμε πρώτα την εισηγήτριά μας την κυρία Βέμπερ, κατόπιν τον κύριο Σόιερ, κατόπιν τον κύριο Τεγκράφ, και κατόπιν να δώσουμε το λόγο στους βουλευτές που θέλουν να ε, πάρουν το λόγο. Παρακαλώ κυρία Βέμπερ, έχετε το λόγο. think it's fair to admit that... Θα πρέπει να πούμε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλά ψηφίσματα σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε πολλά κράτη και στις συζητήσεις προέκυψε ότι τα προβλήματα που εντοπίσαμε σε κάποιες χώρες είναι προβλήματα τα οποία απαντώνται περισσότερο ή λιγότερο σε όλα τα κράτη-μέλη της θα πρέπει ε, φυσικά να παραδοθούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, έχει εκδώσει ένα σημαντικό αριθμό συστάσεων για τα μέσα ενημέρωσης, το ρόλο αυτών, ε, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, κάτι το οποίο είναι και φυσιολογικό, διότι η σημασία των μέσων ενημέρωσης αυτές, αυτή την περίοδο είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι πριν από 20, ακόμα και 10 χρόνια. Σε αυτό το στάδιο θα ήθελα να πω μερικά λόγια για αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Ξεκίνησε με βάση τις συζητήσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια περί της καταστάσεως ε, ε, τις οποίες αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από το γεγονός ότι ο ε, χάρτη των θεμελιωδικαιωμάτων δικαιωμάτων ε, είναι δεσμευτικός τώρα στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε λοιπόν να υπογραμμίσουμε τα άρθρα 11 της Ευρωπαϊκής Χάρτης για την ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης το οποίο αναφέρει ότι όλοι έχουν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης ε, ελεύθερη στην πεποίθηση και να δέχονται να λαμβάνουν πληροφορίες ε, άνευ κανέναν περιορισμό και εγώ με παράδειγμα λέει ότι ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται σεβαστός. Φυσικά ξετάζοντας την έκθεση κάποια ερωτήματα μας έρχονται στο νου. Ποιος θα είναι ο ρόλος των δημοσίων αργών όταν πρόκειται για περιορισμό αυτών των δικαιωμάτων αλλά και για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Τι σημαίνει πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης και η ελευθερία αυτών Αυτή η ελευθερία είναι απόλυτη ή έχει κάποιους περιορισμούς ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωση και τα δημόσια μέσα ενημέρωση ε, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά του. Ε, τι εννοούμε. Θέλουμε να υπάρχει κρατική να υπάρχουν κρατικές ε, ρυθμίσεις, δηλαδή και διευθετήσεις ή θα πρέπει να υπάρχει αυτορύθμιση των μέσων ενημέρωσης. Όλα τα ερωτήματα αυτά λοιπόν χρειάζεται να εξεταστούν μέσα από την έκθεσή μας αλλά έχουμε μια διαδικασία σε εξέλιξη. Αυτή τη... Τώρα είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν Σήμερα προτιμώ να την δίκο νους στους προσεγκλισμένους μας να ακούσω και τους ε, συναδέλφους ε, μέλη της Επιτροπής μας και θα επανέλθω το συντομότερο με ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα και ίσως ε, να συντάξω και ένα αρχικό έγγραφο, ένα πρόχειρο έγγραφο, προτού να περάσω στην τελική σύνταξη της έκθεσης ε, θα... και υποθέτω ότι θα ψηφίσουμε την έκθεση στα τέλη του έτους όταν ε, θα έχουμε και την έκθεση που εκπονεί η ΑΦΕΤ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης Παγκοσμίως Εδώ λοιπόν ολοκληρώνω την παρουσίασή μου και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα ακούσω τους προσκεκλημένους. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Βέμπερ. Σειρά του κυρίου Σόγερ για να μας παρουσιάσει το έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ελευθερία των Άσων Ενημέρωση. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ, τον έχετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τα ευγενικά λόγια που απέφθηνε προς εμάς και για την εισαγωγή που έκανε. Πράγματι έχουμε προσκληθεί στην συνεδρίασή σας ως εμπειρογνώμονες. Μου ζητήθηκε να μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα, στα γερμανικά, Απλά θα ήθελα να σας προειδοποιήσω, γι' αυτό μίλησα αγγλικά, για να βάλετε και τα ακουστικά σας και θα αλλάξω γλώσσα εγώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια σημεία από αυτά που ακούσαμε σήμερα. Ε, μετά την συνεδρίαση θα λάβετε τα τις ε, σχετικές ε, διαφάνειες. Θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω κάποια στοιχεία στο χρονικό διάστημα που μου δίνετε σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο... στα στους λόγους και στο αντικείμενο της μελέτης και κατόπιν θα σας παρουσιάσω τι προσέγγιση επιλέξαμε για να ε, χειριστούμε το θέμα αυτό. Έτσι πιστεύουμε ότι μπορεί η μελέτη μας να αποτελέσει καλή βάση για την ε, έκθεση. Η κυρία Βέμπερ ήδη αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Το 2004 ε, δημοσιεύθηκε μία μελέτη η οποία ανατέθηκε από την ΛΥΜΠΕ τότε ανατέθηκε σαν οργανισμό στο Düsseldorf ε, και ε, ο λόγος για την ανάθεση της μελέτης αυτής ε, ήταν ότι κάποια κράτη-μέλη είχαν εκφράσει ανησυχίες απέναντι στο Κοινοβούλιο υπήρχε Υπήρχαν δύο ψηφίσματα, ένα για την ε, συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, και ένα για την κατάσταση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τον Απρίλιο του 2004 υιοθετήθηκε ψήφισμα από το Κοινοβούλιο και είχε τίτλο για τους σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Ιταλία της ελευθερίας Έκφραση ε, και πληροφόρηση ε, σύμφωνα με το άρθρο 11.2 ε, του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτή ήταν η μελέτη τότε. Σήμερα ζητήθηκε από εμά να επικαιροποιήσουμε την μελέτη αυτή και να λάβουμε υπόψη μας και να εξετάσουμε και την κατάσταση σε νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα που θα αναφέρω πολύ σύντομα. Ε, ε, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας ότι έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, διότι περιέχει δεσμευτικές διατάξεις σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αναφερθώ όμως και στις εξελίξεις που είδαμε μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης μελέτης του 2004. Το 2007 ε, υιοθετήθηκε οδηγία για τις ε, υπηρεσίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, καθώς είχαμε και πρόταση σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε σχέση με τα, το καθεστώς ενίσχυσης. Με το τέλος της χρονιάς του 2010, το φθινόπωρο του 2010, Είδαμε αυτό που προσεκτικά θα ήθελα να ε, περιγράψω ως η περίπτωση της Ουγγαρίας. Ε, αρχές του 2011 είχαμε θέσει σε ισχύ ε, νόμων και ανάλογες αντιδράσεις από την Κομισιόν Γενάρη και Φλεβάρη. Ήδη τον Δεκέμβριο του 2010 είχαμε αντιδράσεις ε, είχαμε ένα ε, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, πέρσι τον Μάρτιο, όπου το Κοινοβούλιο εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το αν οι εθνικές ουγγρικές διατάξεις ανταποκρίνονται στο κοινοτικό κεκτημένο και στις υποχρεώσεις των κρατών μελών να διασφαλίζουν την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την ελευθερία έκφρασης. Τι είναι η βάση για τη δουλειά μας. Ε, πολύ σύντομα όσον αφορά την ε, κατάσταση των πραγμάτων. Στις 15 Φεβρουαρίου είχαμε, στείλαμε την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση στην γραμματεία ΛΥΜΠΕ. Στην διάμεση αυτή έκθεση συμπεριλάβαμε μια σειρά ε, κρατών μελών, ε, τις βλέπετε εδώ πέρα, Βουλγαρία, Τσεχία, ε, Λιθουανία, Μάλτα και Σλοβακία και Γαλλία. Από ό,τι γνωρίζω διατίθεται η έκθεση αυτή. Και αυτή τη στιγμή λαμβάνουμε εκθέσεις από τις υπόλοιπες χώρες. Ε, τι εννοώ όταν μιλώ για εκθέσεις χωρών. Πρόκειται για εκθέσεις ε, εκπονημένες από εμπειρογνώμονες ε, στα κράτη-μέλη, από τους οποίους ζητήσαμε να εξετάσουν συγκεκριμένε στοιχείες με βάση ένα ερωτηματολόγιο που τους στείλαμε σχετικά με τις εθνικές διατάξεις και την εθνική πρακτική όσον αφορά την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωση. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πώς ε, διαμορφώνεται το Σύνταγμα στα διάφορα κράτη-μέλη και όχι μόνο να εξετάσουμε την ε, ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ε, αλλά σημαντική είναι και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των, αρχών, των ρυθμιστικών αρχών για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τέλος, σε μια ε, μελέτη που θα, μια πτυχή που θα μελετήσουμε είναι αν υπάρχουν ε, ε, ρυθμίσεις σχετικά με την υποχρέωση σε κάποιων βασικών υπηρεσιών. Υπάρχει, για παράδειγμα, η υποχρέωση για τα κρατικά κανάλια να παρέχουν ε, κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες, κάποια συγκεκριμένα στοιχεία στους πολίτες. Αντιστρόφως, ε, υπάρχει δικαίωμα των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Έτσι εξετάζουμε τη συνταγματική πτυχή και πέρα από το δίκαιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε και ε, κώδικες δεοντολογίας όπως για παράδειγμα των εφημερίδων, ε, των καναλιών, των δημοσιογράφων. Εξετάζουμε και τους κώδικες δεοντολογίας αυτούς. Σημαντικό είναι Ε, να εξετάζουμε όσον αφορά την ε, ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ε, να εξετάζουμε πόσο ελεύθερα είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παρέχουν πληροφορίες προς τους πολίτες. Και η δεύτερη προσέγγιση είναι πόσο ελεύθερη είναι η πρόσβαση των πολιτών στα, στις πληροφορίες. Θα πρέπει να εξεταστούν και οι δύο αυτές ε, για να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Ε, για παράδειγμα, όσον αφορά την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ε, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην αγορά, ε, τι άδειε προβλέπονται, πώς διαμορφώνεται η ίδια η δουλειά τους, τι περιορισμοί υπάρχουν, τι συγκεκριμένες υποχρεώσεις υπάρχουν για τους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών να διαθέτουν συγκεκριμένο υλικό και επίσης τι δυνατότητες υπάρχουν ε, ε, για τα κανάλια, για τις εφημερίδες ε, να παρέχουν τις πληροφορίες τους προς τους πολίτες. Για παράδειγμα υπάρχει η υποχρέωση να να ε, παρέχονται κάποιες πληροφορίες μέσω καλωδιακής τηλεόρασης, ώστε να είναι ε, προσβάσιμη από όλους. Αυτή είναι η πλευρά της προσφοράς από την πλευρά της ζήτησης. Μας ε, ενδιαφέρει το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες στα διάφορα κράτη-μέλη, το πώς διαμορφώνεται. Και εάν υπάρχει για τους πολίτες δυνατότητα συμμετοχής, δυνατότητα επιρροής, να Μπορούν να πούνε δηλαδή τι είδου πληροφορίε, πιστεύουν ότι θα πρέπει να παρέχονται και πώ. απο Από κάποια κράτη-μέλη υπάρχει συμμετοχή κάποιων κοινωνικών ομάδων ε, όπως ε, για παράδειγμα ε, των Συμβουλίων Ρύθμισης των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει ε, και συνηγόρος του πολίτη, η διαμεσολαβητής για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε κάποια κράτη-μέλη. Υπάρχει εδώ ε, η δυνατότητα των πολιτών να παίρνουν θέση σχετικά με το τι υλικό θα πρέπει να παρέχεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα αν θα πρέπει να παρέχεται μέσω των κλασικών μέσων ή διαδικτυακά ή και διαδικτυακά. Όπως ε, και στη μελέτη του 2004 θα υπάρξει και στη νέα μελέτη ένα κεφάλαιο που εξετάζει ε, ανάλογα με τη χώρα την κατάσταση της ε, αγοράς. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες ε, στον τομέα της τηλεόρασης, της ραδιοφωνίας κλπ. Και επίσης ε, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε και την κατανομή των εσόδων από την διαφήμιση στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τέλος, ζητήσαμε από τους ε, δημοσιογράφους ε, να μας ε, πούν ποιες αλλαγές πιστεύουν ότι είναι απαραίτητες για να λυθούν προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Ε, από ό,τι γνωρίζω αυτό το θέμα, τα προβλήματα ε, έχουν κυρίως να κάνουν με τη συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με την προστασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ε, αυτό έχει να κάνει με την προστασία των πηγών τους, την προστασία δηλαδή από δημοσίευση των πηγών τους και το θέμα της διαφάνειας. Οι πολίτες σε πολλές χώρες φαίνεται να ε, δυσκολεύονται να διαπιστώσουν ποιος είναι ιδιοκτήτης ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης, τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από κάθε δημοσίευση και αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο ε, ασχολούνται ε, αρκετά κράτη-μέλη. Φαίνεται όμως ότι η εφαρμογή των κανόνων δεν λειτουργεί πάντα πολύ καλά στην πράξη. Στην ε, μελέτη θα υπάρξει και ένα ε, άλλο τμήμα, αλλά εδώ θα είμαι σύντομος διότι η κυρία Βέμπερ αναφέρθηκε σε αυτό. Ε, το θέμα του τι περιμένουμε από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Έχουμε κυρίως το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε και συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης Έχουμε επίσης το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην ε, συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε για παράδειγμα τα άρθρα 2 6 που έχουν να κάνουν ιδιαίτερα με τους στόχους και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο άρθρο 11, όπως ήδη αναφέραμε, υπάρχει ε, η ελευθερία της έκφρασης και ο πλουραλισμός και έχουμε τις βασικές ελευθερίες την, ε, τον, ε, την πολιτική ανταγωνισμού και την ε, πολιτική πολιτισμού και επίσης έχουμε και το δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο. Και τέλος, σε μια συγκριτική ανάλυση στο τέλος θα εξετάσουμε και τη σχέση ανάμεσα στα διάφορα κατημέλη καθώς ε, και το επίπεδο των, ε, της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, στα διάφορα κατημέλη και πώς ανταποκρίνονται αυτά στα ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να μπορούμε στο τέλος να δώσουμε κάποιες συστάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα που είναι απαραίτητο να γίνουν. Πληροφορίες σχετικά με τα επόμενα βήματα, πολύ σύντομα προβλέπεται σχέδιο της έκθεσης τέλη Μαΐου και μετά θα έχουμε ένα διάστημα 6 έως 8 εβδομάδων για να ε, συμπεριλάβουμε περαιτέρω επιθυμίες στην έκθεση και στο τέλος θα ολοκληρωθεί η έκθεση αυτή. Ε, ευχαριστώ, θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Να σας υπενθυμίσω ότι στις 11 ε, παρατέταρτο προβλέπεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα αρχίσουν να μπαίνουν ε, πάρα πολλοί συνάδελφοι, τρέχοντας κιόλας, για να ψηφίσουν, γιατί μετά έχουν άλλες υποχρεώσεις. Άρα θα πρέπει μέχρι τότε να έχουμε ολοκληρώσει και έχουμε κι άλλη μια παρουσίαση από τον κύριο Ντεγκράφ, Γκέρχαρτ Ντεγκράφ, ο διευθυντής της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ για, την, ε, για τα μέσα ενημέρωση στον οπτικοακουστικό τομέα. Ίσως καλό θα ήταν να σας δώσω αμέσω κύριε Ντεγκράφ το λόγο και μετά να περάσουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Εισηγήτρια, αγαπητή κυρία Βέμπερ και κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο για να μην καθυστερήσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να κάνω λίγα σχόλια, εισαγωγικό το πρώτο ε, και ουσιαστικά είναι για να σας πω ότι χαιρετίζω την ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η έκθεση της κυρίας Βέμπερ που θα ε, δημοσιευθεί αργότερα σε αυτά τα κείμενα, σε αυτές τις προσπάθειες. Ξέρετε ότι είμαστε και εμείς δεσμευμένοι υπέρ της ε, πολυμορφίας των μέσων, της ελευθερίας του τύπου, είναι αρχές ε, που βρίσκονται στην καρδιά μιας δημοκρατικής και πλουραλιστικής κοινωνίας. Για περί αυτού, άλλωστε, πρόκειται. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να πω ότι επειδή συζητούμε όλα αυτά τα θέματα, ήθελα να πω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ενεργήσει μόνο στο πλαίσιο ε, των αρμοδιοτήτων που τις εκχωρούν οι συνθήκες. Αυτό σημαίνει πολύ συγκεκριμένο ότι σε ό,τι αφορά το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και με βάση το άρθρο 51, το οποίο επανειλημμένω ακούστηκε σήμερα το πρωί, οι διατάξει του απευθύνονται στα κράτη-μέλη μόνο όταν εφαρμόζεται το νοσιακό δίκαιο. Υπό αυτήν την έννοια οι εξουσίες τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι περιορισμένες σχετικά. Θα ήθελα τώρα να περάσω στι δραστηριότητες που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απάντηση και στο ψήφισμα το οποίο ενέκρινε το Κοινοβούλιο τον ε, προηγούμενο Φεβρουάριο για την Ουγγαρία. Θα ήθελα να τονίσω τρεις δραστηριότητες. Πρώτη, ομάδα υψηλού επίπεδου, ανέφερε τα σχετικά ο κύριος Πρόεδρος, μια ομάδα υψηλού επίπεδου η οποία συγκροτήθηκε κατά το δεύτερο ήμιση της προηγούμενης χρονιάς, έχει ε, συνεδριάσει τρεις φορές ε, στο μεταξύ. Πρόεδρος της ομάδας υψηλού επίπεδου είναι ο πρώην πρόεδρος της Λετωνίας, ο καθηγητής Φράιμπεργκερ και τα άλλα τρία μέλη είναι, ο καθη... η καθηγητής Χέρτα Γκεμέλη, πρώην Υπουργός δικαιοσύνη ε, της Γερμανίας, Λοϊς Μιγγέλ Πεσάδο Μαχούρ και Μπεν Χάμεσλιν, τα άλλα δύο μέλη. Η ομάδα κλείθηκε να εξετάσει τους κινδύνους, κάθε είδους κινδύνου κατά της ε, ελευθερίας και του πλουραλισμού του τύπου και των μέσων ενημέρωσης και τις ε, δυνατές δράσεις που μπορούν να ληφθούν. Ίσως ε, και περαιτέρω δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συντάξει έκθεση λοιπόν για την Κομισιόν με συγκεκριμένες συστάσεις για την προστασία, την προώθηση, σεβασμό της ελευθερίας και των και τη πολυμορφίας των μέσων ενημέρωση. Αναμένουμε την έκθεση μέχρι τα τέλη του έτου. και βέβαια τα πορίσματα τη έκθεση, τα πορίσματα των εργασιών τη ομάδα θα δημοσιοποιηθούν, θα ενημερωθεί το Κοινοβούλιο. Είναι ανεξάρτητη ομάδα υψηλού δεν λαμβάνει οδηγίες και εντόλε από κανέναν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μόνο υλικοτεχνική υποστήριξη και μέχρι εκεί. Αυτό το οποίο προσπαθεί να πετύχει η ομάδα αυτή είναι να απαντήσει κάποια ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να εντοπίσει ενδεχόμενου περιορισμού τη ελευθερία των ε, τύπων, ακόμη και κρατικέ παρεμβάσει στη θεωρία ή στην πράξη, αν υπάρχει έλεγχος ε, των μέσων, ε, είναι ανεξάρτητες οι ρυθμιστικές αρχές. Προστασία πηγών, επαγγελματικά δικαιώματα του τύπου και των μέσων ενημέρωσης. Υπάρχουν κίνδυνοι, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αυτό όλο που είπα είναι η πρώτη ε, ομάδα ε, θεμάτων που ενδιαφέρουν ε, την ομάδα αυτή και το δεύτερο είναι το media ownership καθώς επίσης και η λογοδοσία, η εμπιστοσύνη των μέσων. Τον Οκτώβριο έγινε η πρώτη συνεδρίαση, έκτοτε υπήρχαν άλλες δύο και η τελευταία πριν από δύο εβδομάδες Στα θέματα της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας του τύπου ε, έχουν έχει δοθεί μεγάλη προσοχή και σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και σε ό,τι αφορά τους δημοσιογράφους, την ανεξαρτησία και επίσης βασιστήκαμε και τονίσαμε πολύ το θέμα των ε, προτύπων και της δεοντολογίας των δημοσιογράφων. Θα διοργανωθούν και ακροάσεις, περαιτέρω ακροάσεις, Τουλάχιστον πέντε συνεδριάσεις προβλέπονται σε διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επόμενους δύο-τρεις μήνες. Θα διοργανωθούν και ακροάσεις ε, με εμπελκόμενους φορείς και ακαδημαϊκούς. Αυτά σε ό,τι αφορά την ομάδα υψηλού επίπεδου. Οι δύο άλλες δραστηριότητες τώρα, σε οποίες θέλω να αναφερθώ είναι συντομία. Πρώτον, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδίω μέσω μια προπαρασκευαστική ενέργεια που εγκρίθηκε πέρυσι Συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο για να έχουμε ένα κέντρο για τον πλουραλισμό και την ε, ελευθερία του τύπου εντός της σχολής του Σούμαν ε, στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, ένα κέντρο το οποίο πλέον είναι επιχειρησιακό και μία από τις πρώτες του εκθέσεις, μία από τι εκθέσει που επεξεργάζεται είναι η έκθεση η οποία έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την πολυμορφία και την ελευθερία του τύπου. Πριν το καλοκαίρι θα είναι έτοιμη σχετική έρευνα, σχετική μελέτη. Τελευταία δραστηριότητα που θέλω να σας αναφέρω. Η αντιπρόεδρος Νίλη Κρούση έχει συγκροτήσει και μια άλλη ομάδα, Media Futures λέγεται. Αυτή η ομάδα εξετάζει τον αντίκτυπο των τεχνολογικών αλλαγών ε, και της επανάστασης του διαδικτύου στο γενικότερο τοπίο των media. Όπως γνωρίζετε, οι αλλαγές σε αυτό το τομέα, ε, στον τομέα αυτό είναι ταχύτατες, είναι ραγδαίες, ο κλάδος, η βιομηχανία αλλάζει με ταχύτητα τους ρυθμούς, υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι πάροχοι κάθε τόσο στην αγορά και όλα αυτά περιορίζουν πάρα πολύ, βάζουν μεγάλο φόρτο και βάρος και ιδίως τον έντυπο τύπο που αναζητεί νέα μοντέλα για να επιβιώσει πολλές φορές. Και φυσικά υπάρχει ένα πολύ σαφές ενδιαφέρον και στόχος να πετύχουμε πρώτον υγιές και διαφοροποιημένο ε, και ανθούν περιβάλλον για τη βιομηχανία των μίντια στην Ευρώπη και δεύτερον πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτική ε, αναφορά, σε ποιοτικές αναφορές. 25 μέλη έχει αυτή η ομάδα. Διάφοροι τομείς συμμετέχουν και εκπροσωπούνται και δημοσιογράφοι περιλαμβάνονται και περιμένουμε την έκθεση πριν το καλοκαίρι μέχρι τα τέλη του Ιουνίου συγκεκριμένα. Και φαντάζομαι ότι και αυτή η έκθεση θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο. Για να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι η ανάγκη για την προστασία και την πρόθεση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης είναι ένα θέμα που όλους μας αφορά στην Ευρώπη. Ίσως να είναι πιο εμφανές σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες σε κάποιες δεδομένες χρονικές στιγμές, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μας στενά και γι' αυτό θέλω να επαναλάβω πόσο πολύτιμη θεωρούμε την ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την προσπάθεια. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεγκράφ. Αρχίζει η συζήτηση. Έχω έναν κατάλογο με έξι ομιλητές. Δεν έχουμε παρά 20 λεπτά, δύο λεπτά ο καθένας λοιπόν. Σίγουρα είναι ένα συναρπαστικό, πάρα πολύ ουσιώδες θέμα, αλλά σας παρακαλώ να είστε σύντομοι, γιατί έτσι θα αποφύγουμε τις ορδές των ε, συναδέλφων που θα έρθουν να ψηφίσουν στι 11 παρά. Ο κύριος Ταβάρης είναι ο πρώτος ομιλητή. Ευχαριστώ. τα μέσα ενημέρωσης ε, είναι ένα θεμελιώδες ε, ζήτημα. Έλεγα ότι είναι ένα από τα θεμέλια της ε, κοινωνίας μας. Οι πολίτες μας ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την προστασία των μέσων ενημέρωσης. Να βάλουμε συνεχώς αναφορές. Επίσης και πολλές μελέτες γίνονται ανά την Ευρώπη. σε πολλές περιπτώσεις ε, είναι κάπως περιορισμένη η δράση μας, διότι και τα μέσα ενημέρωσης και η Ευρώπη έχουν, διανύουν μια κρίση, έχουμε κρίση στον τομέα της δημοσιογραφίας ε, και έτσι έχει προκριθεί μια τάση που τους οδηγεί τους δημοσιογράφους να ενεργούν με τρόπο, θα έλεγα, στα όρια της παρανομίας. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρουν πολύ καλά τι είναι blog, τι είναι επαγγελματικό blog, τι είναι ερασιτεχνικό blog. Το περιβάλλον λοιπόν των μέσων ενημέρωσης νομίζω ότι ε, οδηγεί σήμερα σε μια ε, ξεκάθαρη εφαρμογή της νομοθεσίας Και ε, διαβάζουμε ειδήσει ε, από απανταχού τώρα πια. Δεν ξέρουμε ούτε ποιον είναι το καθεστώς ε, των μέσων η Κομισιόν μας είπε ότι ναι υπάρχουν οι συνθήκες αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει και η αρχή της επικουρικότητας. Είπατε ότι δεσμεύεται από τον χάρτη κατά την εφαρμογή του, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Έχουμε λοιπόν περισσότερο Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προκειμένου να αριθμίζονται αποτελεσματικότερα αυτά τα ζητήματα. Είπατε ότι χρειάζεται μια διάγνωση, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η Κομισιόν δεν εφαρμόζει τα εργαλεία που έχει στην διάθεσή της τα οποία ζήτησε και απέκτησε, αλλά τελικά δεν τα εφαρμόζει. Δεν τα χρησιμοποιεί. Όλοι γνωρίζουμε ότι απαιτείται αυτή η διάγνωση που αναφέρατε πριν από την ψήφιση νέα νομοθεσία. Εντάξει, θα σταματήσω εδώ διότι υπάρχουν πολλοί αγορητέ που θέλουν να λάβουν το λόγο. ο κύριος Σάιερ είπε ότι θα πρέπει να το, το ζήτημα με τους ε, εμπλεκόμενους, ε, με τους ενδιαφερόμενους, μα όλοι είμαστε ενδιαφερόμενοι. Αν θέλουμε λοιπόν ε, δημοκρατία στην Ευρώπη, πρέπει να έχουμε καλά αποτελεσματικά πρότυπα για τα θέματα της ελευθερίας του τύπου. Ένα παράδειγμα. Ένας δημοσιογράφος απολύθηκε από το κρατικό ραδιόφωνο στην Πορτογαλία διότι έκανε ένα σχόλιο το οποίο ήταν αρνητικό όχι για τη δική μας κυβέρνηση αλλά για την κυβέρνηση της Αγκόλας. Βλέπετε λοιπόν ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει και την δημοσιογραφική και θα πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε να, για να δράσουμε. Ο επόμενος ε, συνάδελφος έχει το λόγο. Και εγώ στηρίζω την ιδέα του να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε αυτές τις πτυχές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσία για τον πλουραλισμό, την ελευθερία των μέσων, το δικαίωμα έκφρασης και το όλο πεδίο των μέσων ενημέρωσης. Με πρόσφατα βλέπουμε κάποιες ε, εκτροπές από τα πρότυπα, από τα στάνταρ ε, και βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιες καταστροφικές τάσεις τα λέγαμε. Όντως ε, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα αναφορικά με τα θέματα της συγχώνευσης ε, κάποιων μέσων ημέρων. Έχουν δημιουργηθεί τεράστια, ε, τεράστια όμιλη δημοσιογραφική οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τον κλασικό τους ε, ρόλο. Αυτό το βλέπουμε και στην, στη χώρα μου, την Βουλγαρία. Παρατηρούμε πως ε, εφημερίδες ε, γίνονται πολιτικό εργαλείο και για να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και συχνά οι διοκτήτες αυτών των μέσων ενημέρωσης είναι τραπεζίτες, εφοπλιστές, πάμπλουτοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ε, ενισχύσουν ακόμα περαιτέρω ε, τη θέση τους στην κοινωνία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν βλέπουμε μια τράπεζα η οποία χρηματοδοτεί ένα μέσο ενημέρωσης, τότε παρατηρούμε ότι αυτή η εφημερίδα μπορεί να γίνει όργανο που στηρίζει την κυβέρνηση, αλλά μπορεί και να συμβεί και το αντίθετο. Βλέπουμε λοιπόν καταστάσεις ε, τις οποίες οι πολίτες ε, δεν ε, κατανοούν, δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο οι εφημερίδες ε, στηρίζουν την εξουσία. Και θα ήθελα να προτείνω προς την κυρία Βέμπερ ότι είμαι στη διάθεσή της διότι ξέρω ότι το έργο της είναι πολύ δύσκολο και περίπλοκο και πολύ ευχαρίστω να την βοηθήσω στο ρόλο της. Ακούγονται διάφορα παράπονα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει, μάλλον επιβάλλει την εφαρμογή των κανόνων της Τρίτη αγοράς με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα, αλλά αν μιλάμε για δημοκρατία, ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ανίσχυη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο χάρτης είναι δεσμευτικός για την εφαρμογή και μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσία. Υπάρχει ένα κενό. Το βλέπουμε πολύ συχνά. Αυτή η πρωτοβουλία είναι μια από τι σημαντικότερε που έχουν αναλυφθεί. Πριν την ένταξη είναι σαφή τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Μετά την ένταξη δεν υπάρχουν συγκριτικά κριτήρια, δεν υπάρχουν benchmarks, δεν υπάρχουν τρόποι εφαρμογής και επιβολής άλλων κριτηρίων. Είναι καλές οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής ΛΥΠΕ και του Κοινοβουλίου Αφενός και της Κομισιόν Αφετέρου για αυτές τις ομάδες το Media Futures Forum και την ομάδα υψηλού επίπεδου για τον πλουραλισμό και την ε, ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Έχω μια απορία, δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί τώρα, αλλά για το μέλλον είναι σημαντική. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε συνέργειες μεταξύ αυτών των δύο πρωτοβουλειών της ΛΥΜΠΕ και της Κομισιόν. Μιλήσατε και για τα πανεπιστήμια. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε λοιπόν συνέργειες. Να έχουμε δηλαδή ένα αποτέλεσμα που θα είναι συνεκτικό, όπου θα υπάρχει πρόταση κοινή, ένα καλό θεμέλιο για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση που ανέφερα πριν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόγκς. Είναι της ελευθερίας του τύπου, έχει δύο ε, πρόσωπα, αν θέλετε. Πρώτα απ' όλα την ελευθερία του τύπου από τον κρατικό έλεγχο, είτε υπό τη μορφή περιορισμών, ε, λογοκρισίας, τιμωρίας, ε, και απ' την άλλη η παγόρευση ε, του τι θα λέει, τι θα κάνει ο τύπος. Και βέβαια το δεύτερο είναι η πρόσβαση στα μέσα. Δικαίωμα πρόσβαση που είναι ένα είδο και νομικό περιορισμό, δεν θα επισέλθω σε αυτό όμω. Θα έρθω σε κάποιε θεμελιώδει αρχέ. Ε, τα κρατικά μίντια, ιδίω από το ακουστικό τομέα, θα πρέπει να ελέγχονται από τον νόμο και θα πρέπει να είναι αμερόληπτα. Πάντοτε όμω πρέπει να είναι ελεύθερα από τον έλεγχο τη εκάστοτε κυβέρνηση. Οι εθνικοί οπτικοακουστικοί φορείς δεν θα πρέπει ε, να δέχονται ε, υποδείξεις και να τους παγορεύεται το τι θα λένε, το τι θα παρουσιάζουν. Θα πρέπει να είναι αμερόληπτοι. Τώρα τα έντυπα. Αυτά και αν θα πρέπει να είναι ελεύθερα. Και φυσικά δεν θα πρέπει να παροτρύνουν σε μίσος ή να ε, κάνουν συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτή είναι ο μόνος περιορισμός η κάλυψη της επικαιρότητα πρέπει να είναι ανεξάρτητη, απ' την άλλη μπορούν να υπάρχουν και τα αρθρογραφήματα τα οποία μπορούν να είναι όσο, το, όσο υποκειμενικά επιθυμεί ο συντάκτης. Επαναλαμβάνω ότι αν υπάρχει δικοσυκοφεντική δυσφήμιση ή παρότρινση σε μίσο στη βία, εκεί αυτό είναι το, ο μόνος περιορισμός. Θα πρέπει να δούμε τώρα. Ε, μιλάμε για την Ουγγαρία και για άλλες χώρες. Τι ελευθερία υπάρχει σε άλλες χώρες. Η Ολλανδική κυβέρνηση πιέστηκε να λάβει δράση την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα να φυλακίσει τελικά ε, τους ε, συντάκτες μιας ιστοσελίδας ε, ενός ε, κόμματος. Ε, πώς μπορούμε να τα θέλουμε όλα τελικά. Απ' την άλλη πλευρά Πολλές φορές διώκονται, φυλακίζονται άτομα τα οποία εκφράζουν μη βίες αλλά ίσως αιρετικές, διαφορετικές απόψεις και για κάποια καθημαϊκά ζητήματα. Στη χώρα μου το Ηνωμένο Βασίλειο, το BBC, ε, δίνει ε, λόγο σε πολλά άτομα που εκφράζουν κάποιες απόψεις ε, χωρίς όμως να δίνει βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν, που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις. Επίση, στη γερμανική τηλεόραση πρόσφατα έγινε συζήτηση για το κατά πόσον θα πρέπει να απαγορευτεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα που πριν από κάποια χρόνια προσπάθησε το κράτος να το απαγορεύσει βάσει προκατασκευασμένων όμως ε, στοιχείων. Μόνο τα θύματα ε, του αποκλεισμού και της απαγόρευσης ε, δεν προστατεύονται τελικά. Άρα ναι μεν ελευθερία του τύπου, αλλά όχι για τους αντιφρονούντες, μόνο για αυτούς που στηρίζουν. Λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, η ελευθερία είναι για όλους. Χαιρετίζω τη σημερινή συστήλα κυρία Φέιτζεν. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της ανεξαρτησίας και της ε, ελευθερίας ε, του τύπου και των δημοσιογράφων, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι συζητούμε αυτά τα προβλήματα στον κόσμο των media. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά ζητήματα, ένα ευρύτατο φάσμα Πολιτικέ πιέσει, επιχειρηματικέ πιέσει, τα μίντια, το νέο φαινόμενο πίσω των κοινωνικών μέσων ενημέρωση και πώς επηρεάζουν την ποιότητα τη πληροφορία ιδίω τα έντυπα μέσα. Το ότι δεν υπάρχει πλέον έρευνα δημοσιογραφική. Συζητάμε εδώ και ένα χρόνο περίπου ε, την περίπτωση της Ουγγαρίας, ε, που έχει κρούσει τον κόδωνα ε, του κινδύνου και έχει σημάνει συναγερμό σε πολλές χώρε. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε τον ανεξάρτητο τύπο. Ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι η Ουγγαρία όμως μια μεμονωμένη περίπτωση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε σαφείς ισχυρού μηχανισμούς για την παρακολούθηση της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε πιο προσεκτικά ε, αυτά που γίνονται στις χώρες μας. Χαίρομαι που ακολούθησε τη σύστασή μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτείνει ένα έδος μηχανισμού για την αντιμετώπιση και την γεφύρωση των χασμάτων που υπάρχουν στην νομοθεσία για τα μίντια. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ε, ανοιχτή, διαφανής η συζήτηση που θα γίνεται στις ε, χώρες μας. Οι δημοσιογράφοι, οι εμπειρογνώμονες να συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο. Συχνά αυτό δεν συμβαίνει. Το είδαμε ξεκάθαρα στην Ουγγαρία. Κάτι άλλο σημαντικό, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, είναι ότι οι κυβερνήσεις και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να αποφύγουν να νομοθετούν για ζητήματα τα οποία αφορούν το περιεχόμενο της δημοσιογραφίας. Θα πρέπει να προωθούν την αυτορύθμιση και να αποτρέπουν, να ε, παρεμποδίζουν οποιαδήποτε πολιτική πίεση. Βλέπουμε διάφορες μορφές ε, πίεσης, εκβιασμού, εκφοβισμού, παράσκησης βίας, ε, πρόσβασης υπηρεσίες. Δεν είναι πάντοτε εύκολο για τους δημοσιογράφους. Αλλά οι δημοσιογράφοι είναι και μια ασφαλιστική δικλίδα κατά της κατάχρησης εξουσίας. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η οικονομική κατάσταση δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου τα μέσα ενημέρωσης εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις επενδύσεις, από την ιδιοκτησία, το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και ένα άλλο θέμα που με ανησυχεί ενδιαίτερα εμένα είναι ότι πάβει να υπάρχει δημοσιογραφική έρευνα. Και στην έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και γενικότερα θα πρέπει να μας απασχολήσουν όλα αυτά τα θέματα. Επίσης, το ψηφιακό περιβάλλον. Πρέπει να το σχολιάσουμε, γιατί μπορεί να ωφελήσει μεν, αλλά την πρόκληση αυτά πρέπει να την αξιοποιήσουμε με το σωστό τρόπο και θα πρέπει να προσαρμόσουμε στις ε, αιτήσει, στα αιτήματα της κοινή γνώμης, στη στρατηγική για τα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε τις νέες αυτές τεχνολογίες, τα νέα εργαλεία ενημέρωσης και πρόσβαση στις πληροφορίες. Επηρεάζεται ο έντυπος τύπος, ο παραδοσιακός έντυπος τύπος. Ακούω ότι στη Βρετανία οι νέοι δεν αγοράζουν καν εφημερίδες, δεν διαβάζουν πια εφημερίδες. Έχουμε το ίντερνετ. Πολλές νέες προκλήσεις λοιπόν. Όλες αυτές θα πρέπει κάπως να τις ε, αντιμετωπίσουμε. Με τα χαράς να συνεργαστώ λοιπόν και εγώ με τη Ρενάτε και με τους λοιπούς συναδέλφους για να εξασφαλίσουμε σε όλα τα κράτη-μέλη την ελευθερία και ανεξαρτησία του τύπου. Πρόεδρος, η εισηγήτρια κυρία Βέμπερ, σύντομα παρακαλώ. Και οι υπόλοιποι να είναι ε, παρακαλώ σιωπηλοί και ήσυχοι. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επικροτώ τη συζήτηση αυτή και τη δυνατότητα να εξετάσουμε την ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα είναι σημαντικό θέμα, το, θέμα για όλου μα και είμαι βέβαιη ότι η κυρία Βέμπερ θα κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω στην έκθεση αυτή. Μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Μέρος ε, του λόγου που ε, έχουμε ασχοληθεί τόσο με το θέμα είναι η Ουγγαρία, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό να μας δώσει την ευκαιρία να επιδείξουμε μια απόλυτα δίκαιη προσέγγιση, ώστε η Ουγγαρία να μην νιώθει ότι ε, την κατηγορούμε άδικα. Σημαντικό είναι να επικεντρωθούμε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση αυτή και αυτή η διαδικασία μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε ακριβώς αυτό. Η ερώτησή μου είναι πώς μπορούμε να εξετάσουμε την ευθύνη καθώς και την ε, ελευθερία ε, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μου γίνεται έρευνα, την έρευνα Λέβινσον, που εξετάζει ε, την κουλτούρα και την ηθική του βρετανικού τύπου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο τύπος μπορεί να καταχρηστεί τις ελευθερίες του και να δημοσιεύει κουτσομπολιά, ε, ε, πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτική ζωή ανθρώπων, ε, κάτι που δεν, έχει να, που δεν αποτελεί είδηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα την εισηγήτρια την κυρία Βέμπερ για να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που συνέβαλαν στη συζήτηση αυτή. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους ε, προσκεκλημένους μας ε, και θα ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω ε, το εξής. Η ενδιάμεση έκθεση σύντομα με τη σύμβαση είναι εμπιστευτική, γι' αυτό δεν έχει διανεμηθεί στους βουλευτές της Επιτροπής ΛΥΜΕ αλλά ε, περιμένουμε να λάβουμε την οριστική σας έκθεση στα τέλη του Μαΐου. Και όπως ήδη είπα, θα σας ενημερώσω όσο γίνεται πιο σύντομα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και θα οργανώσουμε συναντήσεις όχι μόνο με τους κοιόδης εισηγητές ε, αλλά και με ε, τους σημερινούς ομιλητές για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βέμπερ που ήσασταν τόσο σύντομοι ε, κατά την σύνοψη της ε, συζήτησης ε, που μόλις είχαμε. Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστούμε και τους προσκεκλημένους μας, τον κύριο Τεγκράφ και τον κύριο Σόγερ για τις ε, παρεμβάσεις τους. Η γραπτή ε, παρουσίαση ε, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ε, Δικαίου για τα μέσα βασική ενημέρωση θα διανεμηθεί εν ευθέτω χρόνο σε όλα τα μέλη τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Θα ήθελα να σα ε, θυμίσω ε, να έχετε έτοιμη την ε, ηλεκτρονική σα κάρτα. Εάν είσαστε όλοι έτοιμοι, ελπίζω να είστε όλοι έτοιμοι. Εάν όχι, σα παρακαλώ ή βρείτε κάποιον να σας τη βρει ή ενημερώστε μας έχουμε ε, κάποιες ψηφοφορίες, δεν νομίζω ότι θα μας πάρουν πολύ χρόνο. Σας παρακαλώ όμως προσέξτε με. Θα είναι πιο εύκολο για όλους μας να προχωρήσουμε στο, στο, στη συνέχεια της ημερήσιας διάταξης εάν ολοκληρώσουμε τι ε, ηλεκτρονικέ πληροφορίε. Η πρώτη έχει να κάνει με την ε, προστασία των ε, κριτικών υποδομών, επιτεύγματα και επόμενα βήματα προ την παγκόσμια κυβερνοασφάλεια. Συντάκτρια της νομοδότησης είναι η κυρία Άγνες Χάνκης και θα ξεκινήσουμε με αυτή την πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη θα είναι πιο απλή, παρακαλώ συγκεντρωθούμε. Προχωράμε λοιπόν. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κάποιε καταπίπτουν. Προχωράμε στην τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Η 8 καταπίπτει. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κάποιες καταπίπτουν, προχωράμε στη 15 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται, 16 υπέρ. Παρακαλώ.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 λήξη της ψηφοφορίας. Έχουμε 24, 45 υπέρ, δύο αποχές, κανείς κατά. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε ε, την κυρία Χάνκης. Και προχωράμε τώρα στην επόμενη έκθεση, στη δεύτερη έκθεση, η οποία είναι πολύ πιο απλή διότι ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα του εισηγητού μας ε, κυρίου Ταβάρης. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, λίγα λόγια να ευχαριστήσω όλους ε, τους εσκιώδεις εισηγητές ε, και τους συναδέλφους που εργάστηκαν πάνω στο θέμα αυτό. Όπως φαίνεται ότι φτάσαμε στο τέλος της διαδικασίας συναπόφασης, θα ήθελα να σας πω όμως ότι την προηγούμενη εβδομάδα λάβαμε την ε, λυπηρή είδηση ότι ο συνάδελφος από την Επιτροπή που έχει εργαστεί πάνω στο θέμα αυτό τα τελευταία δύο χρόνια πέθανε. Είχε πολλούς φίλους ε, στην Κομισιόν και στο ε, Κοινοβούλιο και θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την ψηφοφορία στην, στη μνήμη της. Σας ευχαριστώ που, για την παρατήρησή σας αυτή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μόλις μάθαμε ότι η κυρία Στεφανία Πασκουέτη απεβίωσε ξαφνικά Είναι πολύ θλιβερό αυτό και θα θέλαμε να τιμήσουμε τη μνήμη της. Θα παρακαλούσαμε να γραφεί στα πρακτικά της, ε, των εργασιών της Επιτροπής ε, ΛΥΠΕ ότι εκφράζουμε την, ε, τα συλληπτήριά μας στην οικογένειά της και στους κοντινούς της. Θα λείψει σε όλους μας. Αφιερώνουμε λοιπόν την έκθεση αυτή στη μνήμη της και προχωράμε στην ψηφοφορία, ηλεκτρονικός έλεγχος για το νομοθετικό ψήφισμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 44 υπέρ, καμία αποχή, 3 κατά. Εγκρίνεται η, ε, το, ψήφισμα, συγχαίρουμε την ε, κυρία Χάνκης και τον κύριο Ταβάρες, σε λήξη των ψηφοφοριών. Προχωράμε στα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης. We're moving on now to point number 13. Περνάμε στο επόμενο σημείο, υπαριθμών 13, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, σημείο 14. Πρόκειται την ενίσχυση της αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του ασύλου εισηγητής ο συνάδελφος κύριος Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Ας ακούσουμε πρώτα την Κομισιόν και μετά θα περάσουμε στην πρώτη ενταλλαγή απόψεων. Η Κομισιόν ενέκρινε μια ανακοίνωση για την ενίσχυση της ελεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του ασύλου προκειμένου να υπάρξει καλύτερη συνεργασία και εμπιστοσύνη ο εισηγητής μας ε, ε μια λοιπόν πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριος Άνταλμπερτ Τζάντσου εκ μέρους της ευρωπαικης επιτροπης και επειτα θα εχουμε μια πρωτη ανταλλαγη αποψεων ο κυριος Άντελμπερτ τζαντσου εκ μερους της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Thank ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση προκειμένου να σας παρουσιάσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Είναι ένα ζωτική σημασία ε, ζήτημα και είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να εγκρίνει μια έκθεση σχετικά με το θέμα. Το ζήτημα της αλληλεγγύης πρόκυψε έντονα πέρυσι, όχι μόνο λόγω των γεγονότων στο Νότιο Μεσόγειο και τις επιπτώσεις αυτών, αλλά και λόγω των πιέσεων που έγιναν προς το ε, σύστημα ασύλου της Ελλάδας. Το αλληλεγγύη ήταν ένα κεντρικό ζήτημα για την πολιτική ασύλου, αλλά για πολύ μεγάλο διάστημα από την απαρχή εδώ και 10 χρόνια από την αντίθεση της πολιτικής. Γι' αυτό λοιπόν η ανακοίνωση της Κομισιόν δεν αποτελεί μόνο αντίδραση στα όσα έγιναν πέρυσι, αλλά ε, βλέπει και πιο στρατηγικά το ζήτημα, πιο μακροπρόθεσμα. Γιατί χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη αλληλεγγύη πρωτοίστως διότι όπως γνωρίζετε τα, ε, οι ροές δεν είναι σταθερές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ετούντων άσυλο, αλλά και επειδή Μολονότι μάλλον ε, αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο πολλές αιτήσει, αλλά αυτές οι αιτήσει δεν είναι τόσο πολλές όσο ήταν στις αρχές της δεκαετίας και δεν είναι τόσο υψηλέ όσο σε άλλες περιοχές του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν είναι ο κατάλληλος χρόνος για να εξετάσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν κάθε απρόβλεπτη ε, ροή. Ε, επειδή λοιπόν οι ροές δεν είναι τόσο υψηλές όσο το παρελθόν, όλα τα αυτά ε, ασκούν πιέσεις διότι είναι ανισόρροπα κατανεμημένες. Ε, παραδείγματος χάρη το πρώτο ήμιση της ε, χρονιάς έξι κράτη έλαβαν περίπου το σύνολο των ετοιμάτων για παροχή ασύλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν φέρει την ευθύνη για να ενισχύσει την αλληλεγγύη ανάμεσα στα κρατημέρια σε θέματα ασύλου και επίσης για να διασφαλίσει ότι όλοι οι τούντες άσυλο ε, γίνονται δεχτοί με αξιο, τρόπο αξιοπρεπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολες και απλές λύσεις και αυτό για δύο λόγους του. Πρώτον, διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό πέραν της αλληλεγγύης στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τις ευθύνες τους σε θέματα παροχής ασύλου και να ε, φροντίζουν τα του οίκου της. Θα πρέπει λοιπόν η λεγή να συνοδεύεται με την ευθύνη, την υπευθυνότητα, δεν μπορεί να αναπληρώσει την ευθύνη των κρατομελών, διαφορετικά το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου θα, ε, θα χρεοκοπήσει. Και, αυτός, και ένας δεύτερος λόγος ε, είναι διότι οι ανάγκη των κρατομελών μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Δεν υπάρχει ένα ε, μια πολιτική κομμένη και ραμμένη για το κάθε κράτος ε, μέλος. Εξαρτάται λοιπόν το πώς αναπτύσσεται κάθε, σε κάθε κράτος το θέμα του ασύλου, αν υπάρχει κατεπίκουσα κατάσταση, κατάσταση, η γεωγραφική θέση της χώρας κλπ. Η ανακοίνωση λοιπόν αυτό το οποίο προτείνει είναι να προσεγγίσουμε την προσέγγιση, να προσεγγίσουμε την αλληλεγγύη για μέσω ανάπτυξης συγκεκριμένων εργαλείων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή με τρόπο ιδιαίτερα στοχευμένο. Αυτό που κάνει λοιπόν η ανακοίνωση είναι να ε, ε, παίρνει την εμπειρία των τελευταίων 10 χρόνων και να την βάλει σε ένα συγκεκριμένο και σαφές πλαίσιο, δηλαδή να δούμε πώς όλα αυτά τα μέτρα λειτουργήσαν και ποια θα πρέπει να είναι η περαιτέρω εξέλιξη αυτών των μέτρων για να τα βελτιώσουμε και να τα συμπεριλάβουμε στο αυτό το, αυτή την εργαλειοθήκη. Έχουμε τέσσερι προτεραιότητε λοιπόν, τέσσερι άξονε αν θέλετε. Πρώτη είναι ε, συνεργασία στην πράξη και τεχνική αρρωγή. Ε, όπως γνωρίζετε υπάρχουν πολλά μέτρα, πολλές συμφωνίες συνεργασίες ανάμεσα στα κρατημέλη αλλά η πρόσφατη σύσταση ε, του ΕΑΣΟ, της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Ασύλου, είναι κάτι το, στο οποίο ελπίζει η Κομισιόν, θεωρεί ότι θα, φέρει μια νέα προσθέμενη αξία και ειδικά ε, με την ύπαρξη του ΙΑΖΟ, μια συνεργασία στην πράξη, στην ουσία, θα γίνει ένας σημαντικός πυλώνας του συστήματος ασύλου. Δεν θα υπάρχουν ε, ε, αυτές οι αρχόκε που υπήρχαν μόνο. Η δεύτερος πυλώνας είναι η, οικονομική ε, αρρωγή και ε, θεωρούμε ότι το Ταμείο Ασύλου ήταν ε, ένα αποτελεσματικό μέσο, μόνο ότι δεν είναι πολύ καλά απεικοδοτημένο, αλλά θεωρούμε ότι μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω αν τα κρατη χρησιμοποιούν ε, τα εθνικά προγράμματα με τρόπο πλέον στρατηγικό για να δημιουργήσουν, να οικοδομήσουν ε, ικανότητες στο σύστημα και ε, δεύτερον θα μπορέσει να ενισχυθεί περαιτέρω από το Ταμείο ασύλου και μετανάστευση. Ε, δεν ε, θα το θίξω το ζήτημα διότι συζητείται σε άλλου χώρου. Η πρόταση τη Κομισιόν περιέχει μια σειρά από χαρακτηριστικά που θα καταστήσουν την χρήση αυτού του ταμείου πολύ πιο ευέλικτη αλλά και πιο στοχευμένη. Ένα ε, άλλο τρίτο άξονα είναι το ζήτημα τη κατανομή των ευθυνών. Ενδεχόμενα αυτό να είναι ένα από τα πλέον ευθύναχα ζητήματα ό,τι φορά την αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν από αυτήν την πρόταση, ε, ε, μάλλον πέραν το τον όρο της κατανομής υπάρχει το ζήτημα το πού βρίσκονται οι αιτούντες έσυλο και ειδικά όσοι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι επικρίνουν τον, ε, το Δουβλίνο, άλλοι που την επενούν. Σε αυτή την ε, περίοδο όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στη μετανάστευση του κανονισμού του Δουβλίνου που πρότεινε η Κομισιόν 2008 και η πρόταση αυτή πρέπει να υιοθετηθεί το 2012 όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα της Στοκόλμης. Επιπλέον της μεταρρύθμισης ε, του κανονισμού του Δουβλίνου σύμφωνα με την απόφαση 2008 θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν συνοδευτικά μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την ε, κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά τα επιπλέον μέτρα με την εθελοντική ε, κατανομή αυτό ε, εμπίπτει από το πρόγραμμα της Μάλτας και η Κομισιόν προτείνει μια μόνιμη ανακατανομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πέραν λοιπόν αυτού του τρίτου άξονα, ειδικά με την ευθύνη, η Κομισιόν θεωρεί ότι το ζήτημα της διακυβέρνησης της διαχείρισης του συστήματος ασύλου με βάση τους μηχανισμούς ε, έγκαιρης προειδοποίησης και αξιολόγησης ε, του ε, κανονισμού του Δουβλίνου, θεωρεί ότι θα μπορούσαν αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουν την συμμόρφωση των κρατών και να υπάρξουν πιο στοχευμένα μέτρα αλληλεγγύης. Η ανακοίνωση λοιπόν εξετάζει αυτούς τους τέσσερις άξονες Το βασικό μήνυμα είναι ότι η Κομισιόν φυσικά και θα διαδραματίσει το ρόλο της για την εφαρμογή όλων αυτών των εργαλείων, αυτών των μέσων, μέσω προτάσεων, αλλά η αλληλεγγύη στον τομέα του ασύλου δεν είναι κάτι που η Κομισιόν από μόνη τη μπορεί να το να πετύχει. Εξαρτάται ιδιαίτερα από τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων, όλων των εμπλεκομένων και ειδικά εξαρτάται από τη βούλη των κρατών μελών να παίξουν το ρόλο τους. Δηλαδή να παρέχουν ε, κονδύλια ε, στην υπηρεσία, να ε, χρησιμοποιήσουν το θέμα της κατανομής σε θελούσια βάση Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν ε, η ανακοίνωση ταυτόχρονα αναγγείλει κάποιες δράσεις της Κομισιόν αλλά και ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους ε, να παίξουν τον ρόλο τους ε, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δράσεις. Όπως τα γνωρίζετε, το Συμβούλιο δέχθηκε την πρόταση της Κομισιόν και ενέκρινε συμπεράσματα σε ένα κοινό πλαίσιο για την αλληλεγγύη στις 8 Μαρτίου. Αυτά τα συμπεράσματα ε, υποστηρίχθηκαν από την Κομισιόν και θεωρούμε ότι επιβεβαιώνουν την ε, δέσμευση των κρατών μελών για την ατζέντα αλληλεγγύης αλλά και ταυτόχρονα τονίζουν το ζήτημα της ευθύνης των κρατών μελών σε ε, ατομική βάση και εξετάζουν επίσης και θέματα ελέγχου συνόρων ασφάλειας κλπ. Λόγω λοιπόν αυτής της ε, εμπλοκής των ενδιαφερομένων είναι ιδιαίτερα σημαντικό το Κοινοβούλιο να προσθέσει τη φωνή του στο ζήτημα και προσβλέπουμε σε μια βοήθεια που μπορούμε να παρέχουμε στο Κοινοβούλιο όπου οπουδήποτε τη χρειαστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ με την Κομισιόν. Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Τρενταφυλλίδη, το συντάκτη της έκθεσης Ιδέας Πρωτοβουλής και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πράγματι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έγγραφο το οποίο παρουσίασε. Θεωρώ σε μεγάλο βαθμό πολύ θετικό το έγγραφο αυτό. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία βέβαια χρήζουν περαιτέρω συζήτηση και υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία θα διευκρινιστούν έτσι περαιτέρω. Μεταξύ των θετικών εξελίξεων που νομίζω ότι έχουν αναφερθεί είναι η ιδιαίτερη μνήμα στην ανάγκη η αλληλεγγύη να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μέτρα. Επίσης, η χρηματοοικονομική αλληλεγγύη με μεγιστοποίηση της χρήση ε, των κονδυλίων, των ταμείων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων με το 2013 και μετά το Ταμείο βέβαια Ασύλου και Μετανάστευσης. Ο ρόλος ε, του ΕΑΣΟ. Πρακτική συνεργασία, τεχνική αρρωγή μέσω του γραφείου, κάτι πάρα πολύ σημαντικό κατανομή επιμερισμός ευθυνών με τη μετεγκατάσταση των δικαιούχων διεθνούς δηλαδή προστασίας. Όλα αυτά τα σημεία θεωρούμε ότι πρέπει να επεκταθούν ακόμη περισσότερο και να αναπτυχθούν ώστε να έχουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες, ε, στην πραγματικότητα του συστήματος ασύλου αλλά και στο σύστημα που θέλουμε να δημιουργήσουμε στο μέλλον. Η εμπειρία, η αξιολόγηση και του σχεδίου μετεγκατάσταση, όπου υπάρχει είναι κάτι πολύ έτοιμο και χρήσιμο. Η ανακοίνωση ε, σχετικά με αυτή τη μετεγκατάσταση είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο όσους χρήζουν διεθνού προστασία, αλλά οι του άσυλο δεν περιλαμβάνονται. Ιδίω όμως όταν γνωρίζουμε ότι αυτό το βάρος, το τανολογικό βάρος, εκεί ακριβώς βρίσκεται. Υπάρχει επίσης η κοινή επεξεργασία των αιτήσεων ε, για την παροχή άσυλου. Αυτό είναι θετικό. Είναι κάτι που προτείνεται και παρότι προς το παρόν είναι αόριστο, είναι ασαφέ και έχει ε, ξεκινήσει μια μελέτη σχετικά, νομίζω ότι πρέπει να εξεταστεί ως ένα μέσο και μέτρο αλληλεγγύη που θα βελτιώσει και την αποτελεσματικότητα. Είναι επίση προφανέ ότι το γραφείο του ΕΑΣΟ ε, είναι ένα γραφείο στο οποίο έχουν εναποτεθεί πολλές ελπίδες και πρέπει να αιτιολογηθεί αυτό. Θα πρέπει να είναι σαφής η εντολή του γραφείου. Και θα πρέπει να δούμε και τι σχέση θα έχει με τον οργανισμό Frontex. Στην σελίδα 4 της ανακοίνωσης Κομισιόν λέγεται ότι Frontex και Άσο θα πρέπει να συνεργάζονται. Και ότι ο Άσο θα πρέπει να ε, θέλει να συμπεριληφθούν οι πτυχές αυτές στις εργασίες της Frontex. Θα ήθελα κάποιε διευκρινήσει από την Κομισιόν. Πρώτη ερώτηση προς την Κομισιόν. Μια αρχή η οποία τονίστηκε και στην παρουσίαση του εκπροσώπου, η αρχή τη αλληλεγγύη και η έννοια του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών. Με βάση το άρθρο 80 της συνθήκης, οι πολιτικές της Ένωσης ε, σε αυτό το άρθρο και η εφαρμογή αυτών θα διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών επιπτώσεων που θα έχουν στα κράτη-μέλη. Όταν λοιπόν καταστεί αυτό απαραίτητο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δρά με συγκεκριμένα μέτρα για να εφαρμοστεί η αρχή αυτή στην πράξη. Ποια είναι η διαφορά σε αυτές τις έννοιε που αναφέρονται. Δηλαδή αλληλεγγύη αφενός, δίκαιο επιμερισμό αυτών αφετέρου. Πώς αυτό επηρεάζει το οποιαδήποτε επιλογή των ενδεχόμενων πολιτικών και των μέτρων τα οποία θα πρέπει να ενταχθούν στον μηχανισμό αλληλεγγύης που εξετάζει η Κομισιόν. Δεύτερο ερώτημα. για του διαφορετικού ε, ετούντε άσυλο που δέχονται τα διάφορα κράτη-μέλη. Το είπε και η Κομισιόν σήμερα το πρωί. Πώ η Κομισιόν βλέπει το ρόλο των κρατών μελών στο πλαίσιο ενό μηχανισμού αλληλεγγύη. Των κρατών μελών λοιπόν που για γεωγραφικού ή άλλου λόγου, ε, δέχονται μικρό αριθμό σχετικά ετούντων άσυλο και προσφύγων. Άρα δεν έχουν μεγάλο φόρτο σε σχέση με άλλες χώρες. Το particular pressure Ιδιαίτερη ε, πίεση, πίεση, massive influx, μαζική εισρωή, είναι έννοιες που τις ακούμε συχνά. Πώς ορίζονται? Ποιος και πώς θα αξιολογήσει την ε, σημασία τους, το νόημά τους. Και έπειτα έχουμε και την έννοια της αλληλεγγύης και την εξισορρόπηση με την ευθύνη, μια άλλη πτυχή της ε, ανακοίνωσης. Αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, τονίζεται μάλιστα και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, και επανειλημμένως έχει αναφερθεί ότι η αλληλεγγύη θα πρέπει να συνοδεύεται από ευθύνη. Υπευθυνότητα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα συστήματά τους μπορούν να ανταποκριθούν στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα δικαίου και θα πρέπει να μπορούν να έχουν τα του οίκους τους του οίκου τους τακτοποιημένα. Αυτό είναι κλειδί για την αλληλεγγύη. Πώς η Κομισιόν βλέπει ακριβώς αυτή την ισορροπία, πώς να αντιλαμβάνεται, ιδίως ό,τι αφορά χώρες που αντιμετωπίζουν ήδη πάρα πολλά προβλήματα στα συστήματα παροχής ασύλου. Η αλληλεγγύη προηγείται, δηλαδή τα μέτρα αλληλεγγύης ή η συμμόρφωση αν δεν υπάρχουν μέτρα αλληλεγγύης, ε, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις ετών. Σε ό,τι αφορά τώρα το πιλωτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης ε, προσφύγων της Μάλτας που έλαβε χώρα το 2011, το μόνο μέχρι στιγμής τέτοιο σύστημα, θα ήθελα να πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αξιολόγηση από την Κομισιόν. Πέραν όμως των κριτικών για το σχετικά μικρό αριθμό των μερών, των τοποθεσιών, φαίνεται ότι ήταν μια θετική εμπειρία. Επίσης αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι η Κομισιόν θα προτείνει ένα εθελοντικό μόνιμο μηχανισμό, αλλά βέβαια με την επιφύλαξη ε, σχετικής μελέτης αντικτύπου. Θα ήθελα να ακούσω κάποια πράγματα και γι' αυτό. Εδώ θα ολοκληρώσω. Θα επανέλθω μετά τη συζήτηση για να σχολιάσω τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ κύριε Τριανταφελίδη. Έχουμε τώρα χρόνο για συζήτηση. Να ξεκινήσουμε την κυρία Γκυγιόμ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακοίνωσή τη, που είναι ιδιαίτερα ποιοτική, και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για τα πρώτα του σχόλια σε σχέση με αυτή την έκθεση πρωτοβουλία. Πάρα πολύ σημαντική έκθεση πρωτοβουλία. Όπω είπα, χαιρετίζω τη σημερινή ανακοίνωση, αλλά θέλω να χαιρετήσω και την ανακοίνωση τη Κομισιόν ε, του Δεκεμβρίου του 2011. Για τρει τουλάχιστον λόγου. Πρώτον, η ανακοίνωση αυτή ουσιαστικά είναι μια αντίδραση ε, σε μια διαπίστωση αποτυχίας, κοινή ε, αποτυχίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι ενεργεί με επικοδομητικό τρόπο, αντιδρώντα σε αυτή την αποτυχία, στην αδυναμία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει με σφαιρικό συνολικό τρόπο τι συνέπειε και τη Αραβική Άνοιξη αλλά και άλλων εσωτερικών φαινομένων. Θα πρέπει να επενθυμίσω ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη αν αντέδρασαν στα πιο πρόσφατα ή παλαιότερα αυτά γεγονότα, δεν ε, το έκαναν όταν χρειάστηκε να υποδεχθούν κάποιου πληθυσμού. Άρα η Επιτροπή στην ανακοινωσή τη βάζει ε, το δάκτυλο από τον τύπο των ήλων και μιλά για αυτή τη συλλογική αποτυχία. Θα ήθελα να χαιρετήσω λοιπόν την ανακοίνωση αυτή, διότι εντάσσεται στο πλαίσιο, ε, σε μια πολιτική ε, κατεύθυνση που αναφέρει την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα ασύλου ως μια αξία. Η αλληλεγγύη είναι πράγματι η θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε. Τρίτο στοιχείο για το οποίο χαιρετίζω την ανακοίνωση. Η προτινόμενη απάντηση είναι μια πλήρη σφαιρική απάντηση. Έχουμε να, ήδη ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση ε, το 2012. Και με την ανακοίνωση αυτή νομίζω ότι μπορούμε έτσι κάπως αποστασιοποιημένα να εκτιμήσουμε τις διάφορες πτυχές αυτής της πολιτικής ασύλου και νομίζω ότι είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος να εξετάσουμε την πολιτική αυτή. Η ανακοίνωση μιλά σίγουρα για κάποιες αρχές που πρέπει να εφαρμοστούν. Και αυτό είναι ο ρόλο τη. Δεν μιλά για τα πολύ πρακτικά ζητήματα. Αλλά σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη, μα παροτρύνει να πάψουμε απλά τα λόγια και να περάσουμε στα έργα. Αυτό μας ζητείτε. Και επειδή σε αυτό το στάδιο μπορούμε και εμείς να εκφράσουμε κάποιους προβληματισμούς μας προς τον εισηγητή, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω ε, τις απόψεις μου και ως κοιόδης εισηγήτρια. Φαντάζομαι ότι η ομάδα μου συμμερίζεται αυτές τις απόψεις. Κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, κάποια βασικά μηνύματα για να αξιοποιήσουμε αυτήν την εργαλειοθήκη που είναι ευέλικτη αλλά κοινή ε, για να βγούμε από το ο καθένας ε, ασχολείται με τα δικά του και για το δικό του συμφέρον. Ένα από τα βασικά μηνύματα που πρέπει να κατευθύνει τη δράση μας είναι τρεις αξίες, τρεις άξονες. Αλληλεγγύη, ε, το ανέφερε και ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Αλληλεγγύη, ευθύνη, επευθυνότητα και αμοιβέ εμπιστοσύνη. Αυτά νομίζω τα περιγράφει και η ανακοίνωση και είναι οι άξονες με του οποίου θα, θα βασιστούμε και θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή. Για τι επόμενε εβδομάδε, λοιπόν θα επεξεργαστούμε αυτό το θέμα. Θέλω να τονίσω και κάτι ακόμα για την οδηγία κατά των διακρίσεων. Το συζητήσαμε και χθε αυτό που θέλω να αναφέρω. Η οικονομική κατάσταση σίγουρα περιπλέκει το έργο που έχουμε να επιτελέσουμε στον τομέα αυτό. Αυτό είναι τη σπάση γνωστό και ξεκάθαρο. Αν έχουμε κοινά εργαλεία, κατά την άποψή μου αυτό θα συμβάλλει στο να μειωθεί το εθνικό κόστος και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το άσυλο, που είναι ένας τομέας στον οποίο οι επενδύσεις ε, για το μέλλον προκαλούν κάποιες εξοικονομήσεις ε, ε, και οικονομικές και σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Δηλαδή βλέπουμε τι μπορούμε να εξοικονομήσουμε, πώς, πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Δεν πρέπει να υπάρξει αδιέξοδο, δεν πρέπει να προσκρούσουμε σε αδιέξοδο για αυτό το θέμα. Αυτή η εργαλειοθήκη λοιπόν πρέπει να είναι ευέλικτη, να είναι λειτουργική, και να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα απτά εργαλεία και μέτρα που θα έχουν επίπτωση ως και ως προς το κόστος. Επειδή γίνεται λόγος και για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αυτή την ε, κοινή πολιτική για το άσυλο, για την αλληλεγγύη, να μην ξεχνάμε και το Συμβούλιο όμως, έτσι, που και αυτό έχει πολύ σημαντικές ευθύνες, γιατί αυτό είναι αυτό που πρέπει να μεταφράσει σε πράξεις και κάποιες πρόσφατες δηλώσεις της 8 Μαρτίου για παράδειγμα για την ε, απτή ε, συγκεκριμένη αλληλεγγύη. Αυτά τα γράφει το Συμβούλιο στο κειμενό του. Τα κράτη-μέλη λοιπόν, το Συμβούλιο ε, καλείται και αυτό. Καλούνται και τα κράτη-μέλη να λάβουν τις ευθύνες τους και να συνεννοηθούν μεταξύ τους σε ό,τι αφορά τα θέματα της αλληλεγγύης για το κοινό πρόγραμμα ασύλου. Σας ευχαριστώ.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 Επιτροπή εκφράζει σαφώς τι εννοεί όταν λέει αλληλεγγύη, τεχνική υποστήριξη, ε, οικονομική αλληλεγγύη, ε, καταμερισμό των ε, υποχρεώσεων και βελτίωση των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Βρίσκω επίσης σημαντικό ότι η Κομισιόν παίρνει σαφή θέση και λέει ότι θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει όπως μέχρι τώρα ε, η οδηγία για την παροχή ε, προσωρινής βοήθειας. Βρίσκω θετικό ότι η Κομισιόν ε, σαφώς δηλώνει ότι ότι η κατάσταση που είδαμε μετά το ότι η κατάσταση που είδαμε ε, το με την ε, Αραβική Άνοιξη δεν ε, έχει καμία σχέση με το Κόσοβο και το 1999. Έτσι. Καθορίζεται η βούληση της Κομισιόν να αντιμετωπίσει τα μεταναστευτικά ρεύματα. Επίση, η Κομισιόν λέει ότι πρέπει να διατηρηθεί το Δουβλίνο, διότι είναι ένα ε, όργανο το οποίο λειτουργεί καλά. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Γίνονται κάποιες συζήτησεις, πρέπει άλλωστε να γίνονται οι συζητήσεις σχετικά με το που υπάρχουν ε, ελλείμματα που, μπορεί, που μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις. Ε, θα πρέπει πάντως να εργαστούμε με αυτή τη βάση. Μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δεν θα πρέπει όμως να ε, αγγίξουμε, να αμφισβητήσουμε την ε, αρχή της πρώτης χώρας εισόδου. Η Κομισιόν δεν θέλει να το αγγίξει αυτό ε, και το Κοινοβούλιο αυτό πιστεύει ότι θα πρέπει να εμείνουμε στον κανονισμό του Δουβλίνου. Επίσης, σημαντικό είναι να υπάρχουν συνοδευτικά μέτρα. Υπάρχει ανάγκη για τέτοια μέτρα, αλλά τα μέτρα αυτά, όπως είναι η κατανομή σε περιπτώσεις επίγουσες, βασίζεται ε, στην αρχή ε, της προαίρεσης ε, του εθελοντισμού και γι' αυτό θα πρέπει να οριστούν οι επίγουσες αυτές περιπτώσεις. Επί της αρχής όμως θα πρέπει Ε, πάντα να αναφερόμαστε στα άτομα που ε, ε, χαίρουν διεθνούς προστασίας. Δεν θα πρέπει να επεκτείνουμε την προστασία όμως σε αυτούς που ζητούν κάπου διεθνή προστασία διότι αυτό αντίκειται σε μια από τις βασικές αρχές που έχουμε μέχρι τώρα. Το θέμα είναι με ε, το Δουβλίνο και με τις δυνατότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή να καταλήγουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε αποφάσεις, ώστε αυτοί που χρειάζονται την προστασία να την λαμβάνουν. Ε, όχι όμως σε αυτούς που δεν δικαιούνται την προστασία. Ε, δεν μπορούμε να ε, κάνουμε ένα άνοιγμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, τέλος, θα ήθελα να σας προειδοποιήσω να μην ξεφύγετε από αυτό που λειτουργεί, από το σύστημα του Δουβλίνου για παράδειγμα. Και αν μία χώρα έχει προβλήματα ή δημιουργεί προβλήματα, δεν θα πρέπει να αλλάξουμε ένα σύστημα που ισχύει και για τα άλλα 26 κράτη. Θα πρέπει να εμείνουμε στο ε, σύστημα αυτό και να ε, παράσουμε βοήθεια όπου είναι απαραίτητη. Να διατηρήσουμε όμως το σύστημα που έχουμε και ε, ναι, ενδεχομένως να βελτιώσουμε το σύστημα όπου έχει ελλείψεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βίξτρομ, σειρά σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, να εκφράσω την εκτίμησή μου για την εξαιρετική δουλειά του κυρίου Τριανταφυλλίδη στο θέμα αυτό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφους για το πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών μας πάνω στι στις εκθέσεις που έχουν να κάνουν με το άσυλο. Ε, η ενδοευρωπαϊκή αλληλεγγύη στον τομέα του ασύλου θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να βασίζεται σε δύο πράγματα, στην ευθύνη και στην αλληλεγγύη. Απαιτούνται και τα δύο για να πετύχουμε τον στόχο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη να εφαρμόζουν τον κανονισμό και να ε, πληρούν ε, τις ε, διατάξεις που έχουν συνυπογράψει. Το σύστημα Δουβλίνο 2 βασίζεται στην ίση μεταχείριση του ετούντος άσυλο σε όλα τα κράτη-μέλη. Σήμερα όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος ε, τον άσυλο ε, κατά 80% έχει πιθανότητες να λάβει άσυλο σε, μία, σε ένα κράτος μέλος και λιγότερο από 1% πιθανότητες σε άλλο κράτος μέλος. Όσο συμβαίνει αυτό, το σύστημα δεν έχει αξιοπιστία ειναι επίση γεγονό γεγονός ότι κάποια κράτη-μέλη δέχονται ισχυρότερη πίεση και δέχονται πολύ περισσότερους ετούντε άσυλο από άλλους. Πρόσφατα ακούσαμε το παράδειγμα του Κωσυφοπεδίου. Να σας δώσω πάλι τα ε, νούμερα από τη Σουηδία. 82.000 άτομα ε, δεχτήκαμε ε, μέσα σε ένα χρόνο και δεν έχουμε εξωτερικά σύνορα. Αν στα σοβαρά ε, θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα κοινό σύστημα θα πρέπει να αναλάβουμε κοινή ευθύνη. Σήμερα 10 κράτη-μέλη λαμβάνουν και ε, δέχονται ε, το 90% των ετούντων άσυλο, το οποίο σημαίνει ότι οι 17 κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να ε, κάνουν περισσότερα και να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες. Ωστόσο, η αλληλεγγύη είναι αμοιβαία. Αλληλεγγύη σημαίνει να πληρεί κανεί τα πρότυπα και να πληρεί τι υποχρεώσει του και, και αυτό είναι σημαντικό για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, να βοηθούν ένα κράτος μέλος το οποίο οποίο ε, υφίσταται ισχυρές πιέσεις. Ε, και τα δύο θα πρέπει να διασφαλίσουμε και η εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντικό θέμα εδώ. Η ε, Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει έλλειψη εμπιστοσύνη. κάτι που δυστυχώ βλέπουμε και στον τομέα του ασύλου. Όταν εξαλείφουμε τα εσωτερικά σύνορα όπω κάναμε, θα πρέπει να ενισχύσουμε, τα... θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη ότι τα εξωτερικά μα σύνορα αποτελούν αντικείμενο σωστή διαχείριση Ναι κύριε Πρόεδρε, απαιτείται εμπιστοσύνη ε, για να διασφαλίσουμε την αλληλεγγύη και χρειάζεται πίστη ε, για να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη. Για την πίστη χρειαζόμαστε αυξημένη αλληλεγγύη. Αυτό αποτελεί τη βάση για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθ' αυτή, όχι μόνο στον τομέα ασύλου και μετανάστευσης. Ε, για μένα είναι σαφές ότι όλοι θα κερδίσουν εάν αυτός ο κύκλος είναι σταθερός. Είναι όμως πολύ εύθραυστος και μπορεί εύκολα να χαλάσει. Όπως ακούσαμε από τον εισηγητή, το άρθρο 8 της συνθήκης ε, εφαρμόζεται στον τομέα ε, αλληλεγγύης και ε, μετανάστευσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ανατρέχουμε συχνότερα στο άρθρο αυτό και να σκεφτούμε τη σημασία του. Οποιαδήποτε μέτρα μπορούμε να λάβουμε για να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη, την εμπιστοσύνη και την πίστη θα ενισχύσουν την ένωσή μας αυτή καθ' αυτή. Εγώ πάντα θα στηρίζω τέτοια μέτρα και γι' αυτό η ανακοίνωση αυτή κατά τη γνώμη μου είναι πολύ θετική. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου πάνω σε ένα κοινό πλαίσιο για πραγματική, πρακτική αλληλεγγύη μεταξύ ε, προς τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν αυξημένη πίεση στο σύστημα ασύλου τους, ε, μεταξύ άλλων μέσω μεικτών μεταναστευτικών ροών, με εξέπληξε πολύ θετικά, διότι υποδεικνύει τη σημασία της ευθύνης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ο ε, και η παράγραφος ε, πάνω στις ε, μετακινήσεις είναι πάρα πολύ σημαντική καθώς και η ε, αναφορά της οδηγίας για την επιστροφή. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει το Συμβούλιο να δείξει ότι παίρνει στα σοβαρά την αλληλεγγύη όπως προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο μας και στην Επιτροπή μας με τις εκθέσεις τις οποίες χειριζόμαστε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Χίρσου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω εισηγήτρια για τους φιλελεύθερους ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την ανακοίνωση αυτή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δεσμευτούμε δούμε ότι θέλουμε έναν ε, κοινό χώρο ε, ε, ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και γι' αυτό το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να ξεφύγουμε. Η αλληλεγγύη και η ευθύνη πάνε χέρι-χέρι κατά τη γνώμη μου και θα πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη που έχουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή των μέτρων αλλά και τα κράτη-μέλη που ε, ίσως ε, είναι πιο επιφυλακτικά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τα παρακινήσουμε ε, να έχουν μια πιο ενεργό πολιτική ασύλου. Πιστεύω ότι και στο πλαίσιο της θεσινής μας συζήτησης ε, για το Ταμείο ε, για τη Μετανάστευση και το Άσυλο ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη νέες πτυχές οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν και κεντρικό θέμα σίγουρα είναι η εφαρμογή, πολύ απλά η εφαρμογή των οδηγιών που ισχύουν για το Άσυλο και των μελλοντικών. Αυτό θα πρέπει να προσέξουμε. Όσον αφορά το Δουβλίνο 2, θα ήθελα καταρχήν να πω ότι φυσικά θα ε, το, το επανεξετάσουμε, θα πρέπει να βελτιωθεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά την κατάσταση. Ε, ο συνάδελφος το είπε ήδη, βρισκόμαστε ε, στη θέση όπου ο απόλυτος αριθμός ε, των ε, ετούντων άσυλο ε, συγκεντρώνεται σε πέντε χώρες μόλις και ε, ο μεγάλος αριθμός των κρατών μελών δεν κάνουν τίποτα παρότι θα υπήρχε η δυνατότητα να δεχθούν ετούντες άσυλο. Εάν, το αποτελ... Εάν αυτό είναι το αποτελέσμα του Δουβλίνου 2, τότε πιστεύω ότι σίγουρα δικαιολογείται να επανεξετάσουμε το Δουβλίνο 2 και να σκεφτούμε μήπως ε, μία δυνατότητα ήταν, θα ήταν οι κλίδες κατανομής. Να εξετάσουμε πόσο πληθυσμό έχει ε, η κάθε χώρα, πόση επικνότητα πληθυσμού. Ε, κατά τη γνώμη μου, Ε, αυτό θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα περισσότερα κράτη-μέλη ε, να συμμετέχουν ε, με αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση του θέματος των ετούντων άσυλο. Δεν πιστεύω ότι πρέπει εκ των προτέρων να αποκλείσουμε τη συζήτηση αυτή θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εθελοντικά προγράμματα ή να υπάρχει συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Θα πρέπει, δηλαδή θέλουμε το Δουβλίνο 2, θα πρέπει όμως ε, να κοιτάξουμε τα αποτελέσματα του Δουβλίνου 2 και να δούμε ε, μήπως υπάρχουν ε, άλλοι τρόποι, άλλοι μηχανισμοί οι οποίοι να είναι πιο αποτελεσματικοί για να πετύχουμε την αλληλεγγύη και την ευθύνη που θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χολμάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ε, επικροτώ το έγγραφο της Κομισιόν. Υπάρχει εδώ πολύ υλικό για συζήτηση. Το γνωρίζουν όλοι αυτοί που ασχολούνται με τις ε, οδηγίες ασύλου εδώ και δυόμιση χρόνια, όπως εγώ. Μερικοί ασχολούνται ακόμα περισσότερα χρόνια με το θέμα αυτό, έχουν ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Νομίζω ότι τα προβλήματα θα μας συνοδεύσουν ε, ε, και κατά τη διάρκεια της εξέτασης αυτού του φακέλου που, μας, ε, που αντιμετωπίζουμε εδώ και δυόμιση χρόνια. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να μπω σε μια γενική συζήτηση, αλλά θα ήθελα να, αναφέρω, να, θέσω τρία ερωτήματα. Το πρώτο, πολύ σωστά αντίθεται, είναι το θέμα της συνεργασίας κατά την εξέταση των αιτήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κάθε κράτος μέλος ε, δεν ε, είναι αρμόδιο. Αλλά, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγή ε, διερμηνέων, για παράδειγμα, διότι για τις μικρές χώρες είναι πολύ δύσκολο να βρουν διερμηνείς για την κάθε περιφερειακή διάλεκτο στην Αφρική. Η Αγγλία, η Γερμανία για παράδειγμα έχουν μεγάλο δυναμικό, η Αυστρία εν μέρη επίσης ε, θα μπορούσε λοιπόν η δυνατότητα αμοιβαίας βοήθειας και συστηματοποίησης της βοήθειας αυτής. Αυτό θα το θεωρούσα πολύ θετικό, διότι από τη μία μεριά εξυπηρετεί τον πρόσφυγα να μπορεί να παρουσιάσει την υπόθεσή του στην ε, την υπόθεσή του, ε, αλλά βοηθάει και την, την λύση των υποθέσεων καθώς και την γρήγορη επεξεργασία των υποθέσεων ώστε ε, αυτοί που δικαιούνται την προστασία να μπορέσουν να ενταχθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα και οι άλλοι να μπορέσουν να επιστραφούν πιο γρήγορα εάν δεν έχουν δικαίωμα παρανομής. Πιστεύω ότι με την συνεργασία αυτή και το θέμα της επιστροφής και ε, της βοήθειας επανεισδοχής ε, στα κράτη-μέλη είναι πολύ σημαντική, διότι μια συγκροτημένη επανεισδοχή είναι σημαντική. Ε, άκουσα Έλληνες ε, υπαλλήλους να μου λένε πόσο δύσκολο είναι να επικοινωνήσουν με άλλες χώρες επειδή οι χώρες ε, αυτές δεν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και που δεν ήθελαν καν να δεχθούν τα αιτήματα, τα ερωτήματα των Ελλήνων υπαλλήλων, πόσο μάλλον να απαντήσουν. Ε, μια τέτοια συνεργασία θα ε, βοηθήσει, θα αυξήσει σίγουρα τη δυνατότητά μας. Ε, τα κράτη-μέλη που θέλουν να εντάξουν στις κοινωνίες τους αυτούς που δικαιούνται προστασία ενδιαφέρονται να υπάρχει και ένας καλός μηχανισμός επιστροφής και επανεισδοχής. Ε, διότι έτσι το κίνητρο ε, να πάει κάνει σε μια χώρα όταν ξέρει ότι δεν έχει, καμία, ε, δεν έχει κανένα δικαίωμα ασύλου θα οι περιπτώσει αυτές θα μειωθούν αν υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός Επίση, Επίσης, ε, το θέμα της Τουρκίας, η πίεση προς την Ελλάδα προέρχεται και από το γεγονός ότι στην ε, περιφέρεια του Εύρου η ε, έλεγχη στα αεροδρόμια όσον αφορά το εμπόριο ανθρώπων και, την, και το οργανωμένο έγκλημα στην Τουρκία δεν θεωρείται ακριβώ προτεραιότητα, για να το πω πολύ ήπια. Ε, αυτό σημαίνει ότι η πίεση προ την Ελλάδα από λαθρομετανάστευση ε, είναι αυξημένη. Ε, δεν έχει εφαρμοστεί το δίκαιο ασύλου όπως προβλεπόταν και γι' αυτό η κατάσταση έχει χειροτερέψει πάρα πολύ. Θα με ενδιαφέρε λοιπόν να μάθω από την Επιτροπή εάν ε, προτίθεται να ασκήσει περισσότερη διπλωματική πίεση στην Τουρκία, ώστε ε, η Ελλάδα ε, και αργότερα και η Βουλγαρία που έχει σύνορα με την Τουρκία να μην υφίστανται ισχυρότερη πίεση θα μπορούσε να παρασχεθεί βοήθεια ε, όσον αφορά την καταπολέμηση της, του εργανομένου εγκλήματος και, του, και, της εμπορίας ανθρώπων. Ευχαριστώ κύριε Σταβάρες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα μιλήσω την μητρική μου γλώσσα. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Τριανταφυλλίδη και να πω ότι μπορεί να βασιστεί στην ομάδα των Πρασίνων κατά την επεξεργασία και κατάρτιση του εγγράφου της. Ε, εισηγητής είναι ο κύριος ε, αλλά μια που ασχολούμε με το θέμα της ε, κατανομής το οποίο σχετίζεται με την επανεγκατάσταση είμαι στη διάθεσή σας ε, όποτε θελήσετε. Εξάλλου είναι και μια εργασία την οποία θα κάνουμε όλοι μαζί στο πλαίσιο των ε, δημοσιονομικών προβλέψεων. Τώρα όπως είπε και η κυρία Βίκστρομ, με ότι κάτι γνώμη μου περιέγραψε απόλυτα καθαρά το, το γεγονός ότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος ε, που λειτουργεί. Πρέπει λοιπόν να αντιστρέψουμε την ε, φορά για να μπούμε σε έναν ε, σε μια κατάσταση πολύ πιο φυσιολογική, πολύ πιο ήρεμη, πολύ πιο ήπια, να μπούμε επιτέλους σε έναν ενάρετο κύκλο ε, ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ετούντων άσυλο στην Ευρώπη. Είμαι διάθεση λοιπόν και κρίνω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του προβλήματος βρίσκεται στο Συμβούλιο. Δεν είδα τόσες χώρες να φοβούνται ε, απέναντι στην ε, έννοια αλληλεγγύη. Ζητήθηκε να υπάρξει προσφυγή στο άρθρο 81 και, αλλά υπόθηκε ότι ναι μεν υπάρχει αυτό το άρθρο, αλλά θα πρέπει ποτέ να προσφύγουμε σε αυτό. Τότε λοιπόν πώς θα υλοποιήσουμε κάποιες πολιτικές ε, αλληλεγγύης ε, ενεργητικές χωρίς να προσφύγουμε σε αυτό το άρθρο. Πρέπει λοιπόν εμείς ως Κοινοβούλιο να κάνουμε μια προσπάθεια διαπαιδαγώγησης θα έλεγα για το ζήτημα αυτό. Τώρα για να καταλήξω λέγοντας τα εξής. υπόθηκε ότι το κανονός του Δουβλίνου δεν αντιμετωπίζει κρίση, αλλά κρίση υπάρχει σε συγκεκριμένε χώρες. Με αυτό γίνεται σε περίπτωση κρίσης. Υπάρχουν κάποια αδύναμη, ε, αδύναμη κρίκη και ε, γι' αυτό μιλάμε για κρίση. Το... Εάν το Λουξεμβούργο είχε κάποια ιδιαίτερα εξωτερικά σύνορα, τα οποία ασκούνται πιέσεις, ε, τότε ήταν και το Λουξεμβούργο μία από τις χώρες ε, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Μπορούμε όμως ε, να σκεφτούμε και κάποια χώρες που έχουν κάποια οικονομικά προβλήματα σοβαρά, π.χ. η Ελλάδα. Να λοιπόν ε, ένα αδύναμο σημείο του κρίκου. Στην Αμερική είχαν εφεύρει την έννοια της απουσίας αδύναμου στοιχείου, αλλά μετά το εγκατέλειψαν. Πάντα υπάρχει κάποιο αδύναμο σημείο, αδύναμο στοιχείο, αρκεί να τα εξετάσουμε, να τα αναλύσουμε και να, θα πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι πρόβλημα και του Δουβλίνου 2 και κάτι ακόμα χρειαζόμαστε μια προσέγγιση η οποία θα βασίζεται στην πραγματικότητα, μια ρεαλιστική προσέγγιση. 80% των προσφύγων ε, ανά τον κόσμο προσπαθούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, μικρότερο φυσικά, το οποίο παραμένει στις ε, χώρες ε, στις οποίες είχε μεταβεί, διότι πέραν της γεωγραφικής εγκύρητας υπάρχουν και κάποια, κάποιες παραδόσεις, κάποια πολιτικά στοιχεία που τους κάνει να επιστρέψουν. Αλλά όταν μιλάμε για πρόσφυγες, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πρόσφυγες οι οποίοι δεν έχουν άλλη δυνατότητα από το να επιστρέψουν στη χώρα τους. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για επιστροφή στο Ιράκ, διότι ορισμένοι επιστρέφοντας στο Ιράκ θέτουν σε κίνδυνο την ζωή τους. Και αυτό το διαπιστώνουμε καθημερινά. Για τη Συρία, παραδείγματο χάρη. Είτε όλα τα χρήματα έχουν δαπανηθεί, είτε πάνε σε λάθο ε, χέρια. Και εάν επιστρέψουν σε, κάθε, σε κάποια αυτές τις χώρες ε, κινδυνεύουν ε, ακόμα και να απαγχωνιστούν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ πιο προσεκτικά το ζήτημα. Thank you. Solidarity is uh, an emotively Κοιτάξτε, η αλληλεγγύη είναι ένας ε, ωραίος ε, όρος. Ε, η συμφωνία θα ήταν καλύτερη, αλλά η συμφωνία δεν πρέπει να είναι αυτόματη. Θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία αφού εξεταστούν αποτελεσματικά το ζήτημα. Υπάρχουν λοιπόν ένας δυσανάλογος αριθμός ετούντων ασύλου, αλλά είναι θύματα ε, παράλογων ε, διευθετήσεων σε ό,τι φορά το άσυλο, τη χορήγηση ασύλου, όπως π.χ. η αρχή τη μη ό ε, για να μην επιστρέψουν σε δίθεν ε, επικίνδυνα κράτη. Πολλοί έρχονται στην Ευρώπη παρακάπτοντας ε, ασφαλείς ε, χώρες. Η Ελληνική σήμερα ορίστηκε ως ε, το σωστό μοίρασμα της ευθύνης. Δεν Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει απόλυτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όσους Λοιπόν, αν είναι να έχουμε αλληλεγγύη, θα πρέπει να ε, πάψουμε να βλέπουμε και εμείς και οι άλλοι την Ευρώπη ως μια Ελλάδα προς άρμεγμα. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν, αν θέλει τώρα να απαντήσει στα σχόλια που ακούστηκαν, προτού να δώσουμε το λόγο κύριο Τριανταφυλλίδη για να κλείσουμε το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά ακούστηκαν πάρα πολλά σχόλια τα περισσότερα των οποίων ήταν ιδιαίτερα εύστοχα. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα που απευθύνθηκε από έναν βουλευτή στην Επιτροπή και δεν θα σχολιάσω τις απόψεις των βουλευτών. Διαφορές μεταξύ αρχή της ε, αλληλεγγύης και αρχής της, ε, του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών. Είναι ερώτηση παγίδα κατά κάποιο τρόπο. Δεν θα σας εξηγήσω τώρα αναλυτικά τις σημειολογικές, μεσιολογικές και φιλοσοφικές διαφορές των ενιών, αλλά νομίζω ότι ο στόχος αυτής της ανακοίνωσης είναι ακριβώς να δείξει με ποιο τρόπο μπορούμε να πετύχουμε την ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών ενιών, δηλαδή της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών. Και νομίζω ότι αυτό σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το μεγάλο ερώτημα τι προηγείται. Προηγείται η αλληλεγγύη ή προηγείται η ευθύνη. Η θέση της Κομισιόν επ' αυτού είναι ότι πηγαίνουν χέρι-χέρι, συμβαδίζουν οι δύο αρχές. Κάποιοι ενδιαφερόμενοι εμπλεκόμενοι φορές θα σας πούνε ότι η αλληλεγγύη έπεται ε, ή προηγείται, εξαρτάται. Αλλά αυτή δεν είναι η θέση της Κομισιόν. Εμείς ε, αυτό που επιδιώκουμε είναι την ισορροπία μεταξύ των δύο ενιών. Ο κύριος ρώτησε πώς βλέπει η Κομισιόν το ρόλο των χωρών μελών που δεν έχουν βάρος μεγάλο, δηλαδή δεν δέχονται πολλές αιτήσει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα ήθελα να πω ότι και σε αυτό το σημείο η άποψη της Επιτροπής στη σχετική ανακοίνωση είναι ότι τα κράτη-μέλη πραγματικά ε, έχουν να παίξουν ένα ρόλο ο ρόλος τους όμως ο βασικός είναι να δημιουργήσουν ε, τις υποδομές στα ίδια τους τα συστήματα για να μπορέσουν στο μέλλον να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες ε, εισρωές επειδή οι μεταναστευτικές εισρωές ε, είναι Σε Αυτή τη στιγμή έχουμε στα νότια σύνορα εισρωές αλλά μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε εισρωές από τα ανατολικά σύνορα. Δεν ξέρω. Άρα θα πρέπει να προωθήσουμε τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών. Και βέβαια τα ευρωπαϊκά ταμεία θα πρέπει να αξιοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο, με στρατηγικό τρόπο δηλαδή. Δεύτερον, αυτά τα κρατημέλη που δεν είναι τόσο βεβαρημένα σίγουρα πρέπει και αυτά να φροντίσουν να παράσχουν την πρακτική υποστήριξη στο πλαίσιο και του ΕΑΣΟ προς τα άλλα κράτη-μέλη. Ένα άλλο πολύ συγκεκριμένο ερώτημα που μετέθη ήταν ο όρος Particular Pressure Mass Influx. Τεχνική όρη, άκρος τεχνική όρη, αλλά έχουν οι όροι αυτοί μια πολύ συγκεκριμένη σημασία στο πλαίσιο των νομικών πράξεων. Η ειδική, ιδιαίτερη πίεση ε, είναι ε, ένα ολόκληρο άρθρο αφιερωμένο σε αυτόν την έννοια, στον κανονισμό του ΕΑΣΟ. Σχετικά χαλαρά βέβαια ορίζεται η έννοια, αλλά υπάρχουν ενδείξεις για το τι πρέπει κανείς να εννοεί ως ιδιαίτερη πίεση. Και σε ό,τι αφορά τη μαζική ροή mass influx, αυτή η έννοια σχετίζεται πάρα πολύ με την οδηγία την προσωρινή προστασία, temporary protection. Πάλι έχουμε ένα συγκεκριμένο ορισμό για την έννοια αυτή που σχετίζεται στενά με την έννοια των εκτοπιστέντων ατόμων που, μπορούν να, ε, που δεν μπορούν μάλλον να γυρίσουν στη χώρα τους λόγω των συνθήκων που επικρατούν εκεί. Ένα άλλο ερώτημα ή μάλλον αίτημα ήταν ε, για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτό το μόνιμο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που παρουσιάζει η Κομισιόν. Εμείς σίγουρα θα αντλήσουμε τα διδάγματα από αυτό το πιλωτικό σχέδιο που είναι ακόμα σε εξέλιξη. Εξού και είναι δύσκολο στην παρούσα φάση να σας πούμε ακριβώς ποια είναι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ποια θα είναι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αυτού του πιλωτικού προγράμματος ε, θα αποτελέσει ένα σημαντικό κομμάτι της μελέτης αντικτύπου για αυτό το μόνιμο πρόγραμμα αντικατάσταση, συνεργασία με τη Μάλτα και με τα άλλα συμμετέχοντα κράτη και με τον Ιάζο. Και ανάλογα με το πώς ε, θα σχεδιαστεί αυτός ο μηχανισμός, σίγουρα θα είναι ένας εντελοντικός μηχανισμός, αυτό το έχουμε αποφασίσει, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει και κάποια σχέση με τους κανόνες που διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευση. Για να δούμε πώς θα χρηματοδοτείται αυτό το σχήμα, αυτός ο μηχανισμός. κυρία Χολμάγερ επίση έθεσε ένα συγκεκριμένο ερώτημα για τον Εύρο και για την Τουρκία. Δεν κατάλαβα ακριβώς το ερώτημα. Δεν ξέρω, ε, ίσως να μην το κατάλαβα καλά εγώ, αλλά αυτό που θέλω να πω Εκτός ε, μικροφώνου το σχολείο της Σω Ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και διμερώς. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την ε, Υπηρεσία εξωτερική δράση συνεργάζεται με την Τουρκία εντατικά για την εφαρμογή της ε, συμφωνίας περί επανιστοχής και φυσικά πρέπει να υπάρξει βοήθεια προς την Ελλάδα για τη βελτίωση του ελληνικού συστήματος παροχής ασύλου. Στην ανακοίνωσή μας ε, υπάρχει ε, ενημέρωση και εμεί σίγουρα είμαστε δεσμευμένοι να βοηθήσουμε την Ελλάδα και από τεχνικής και από οικονομικής πλευράς μέσω του ΙΑΖΟ και άλλων κρατών μελών τεχνικά ενισχύουμε την Ελλάδα όσο μπορούμε. Αυτά ήταν από μένα. Κύριε Τρενταφυλλίδη, ο λόγος σε εσάς. Uh, Κοιτάξτε, είναι περιορισμένος ο χρόνος. Ε, θα περιοριστώ και εγώ ε, ευχαριστώντας την Κομισιόν για τις απαντήσεις που μου έδωσαν, αλλά και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους, Γκυγιόμ, Πέρκελ, Βίλστρομ, Χέρσ, Χοκμάιερ, Ταβάρες, Μπρόγκς, για τις ε, πολύ σημαντικές προτάσεις και συστάσεις θα τα λάβω υπόψη μου. Να πω πως ε, πέραν ε, των σχολείων έλαβα θέσεις και απόψεις από ακαδημαϊκούς κύκλους, από μη κοινωνικές ε, οργανώσεις κλπ. Και θα, ε, θα φροντίσω πριν από τα τέλη Απριλίου να έχουμε την έκθεση, μετά θα ακολουθεί συνεδρίαση με τους σκιώδης ηγητές και προτίθεμαι να, παρα, να υποβάλω την ε, έκθεσή μου στην Επιτροπή τον Ιούλιο και να πάμε στην Ολομέλεια μετά από τις τερνές διακοπές ε, το Σεπτέμβριο δηλαδή. Ευχαριστώ. Προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ κύριε Τριανταφυλλίδη, ευχαριστώ και όλα τα μέλη που έλαβαν μέρος στην ε, συζήτηση κύριος Γιάνξ, ο οποίος ε, μας μίλησε για την θέση της ε, Κομισιόν πριν από την έκθεση πρωτοβουλίας ε, που θα υποβάλουμε στο εγγύς μέλλον. Περνάμε στο επόμενο σημείο της Μεσσίας Δετάξεως, είναι το τελευταίο για σήμερα το πρωί και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά τις 15.00. Περνάμε στο σημείο 15 που αφορά την κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών. Εισηγητής ο κύριος Γιάν Μίλντερ. Σκοπός ε, της συζήτηση είναι η παρουσίαση του θέματος μετά από τον τριμερή διάλογο. Παρακαλώ όσοι αποχωρείτε να το πράτετε ησύχως και να μην ταράζεται το κλίμα. Ας ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γιάν Μιλντερ για την κατάσταση όπως αυτή έχει προκύψει μετά από τον τριμερή διάλογο και να έχουμε υπόψη μας πως υπάρχουν τρία πολιτικά διακυβεύματα. Πρώτον, αδειοδότηση κατά της καταχώρησης. Ε, ανάθεση εξουσιών στην Κομισιόν για να κάνει παραρτήματα και τρίτον ε, η ε, εξαίρεση του αζότου Ευχαριστώ Πρόεδρε. Παρουσιάζω την... Παρουσίασα μάλλον την έκθεσή μου πέρυσι τον Ιούλιο και 15 Ιουλίου είχαμε προθεσμία κατάσταση τροπολογιών. Αυτό σημαίνει ότι χάσαμε ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη μία εβδομάδα αργότερα στην Ορβηγία όπου γνωρίζετε όλοι τα φρικτά συμβάντα. Το λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των ψηφοριών, όπου 49 ψήφισαν υπέρ ε, στους 50, υπέρ των συστάσεων που κάναμε. Ποια ήταν τα βασικά συμπεράσματα λοιπόν. Πρώτον, Κατά την πώληση προδρόμων ουσιών εκρηκτικών, η Κομισιόν πρότεινε ένα σύστημα αδειοδότησης, ε, το οποίο σημαίνει ότι για ορισμένα προϊόντα που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο, αν θέλετε να αγοράσετε ένα από αυτά, μπορείτε, μάλλον πρέπει να έχετε άδεια. 49, όπως σας είπα, από τους 50 υπερψήφισαν. Στην μετέπειτα συζητήσεις με, τον, με το Συμβούλιο, αυτό έλαβε μια αντίθετη θέση. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει ένα σύστημα αδειοδότησης, αδειών, σε άλλα κράτη-μέλη έχει το σύστημα της καταχώρησης και σε άλλα προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σύστημα. Δεν ισχύει τίποτα. Αυτό είναι δύσκολο θέμα. Άλλη διαφορά είναι ότι η Επιτροπή μας θέλει να παραμείνει στην συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου, Κομισιών και Κοινοβούλιο αναφορικά με τις πράξεις ε, κατεξοδότηση. Το Συμβούλιο θέλει να έχουμε μια εξαίρεση μια και προτείνει έναν κατάλογο A και έναν κατάλογο Β στον οποίο συμπεριλαμβάνουν αυτά τα προϊόντα, τις ουσίες. Η ε, Συμβούλιο λοιπόν θέλει μια νέα διαδικασία, εάν πρόκειται να προσθεθούν προ... Ε, ε, ουσίες στον κατάλογο Α ή αν πρόκειται να διαγραφούν. Εμείς όμως είπαμε θέλουμε να παραμείνουμε στην αρχική συμφωνία που είχαν συνάψει τα τρία θεσμικά όργανα. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι το... η αζωτούχος αμμονία έχει είχε διαγραφεί και εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τηρήσει αυτή Αυτό το νητρικό αμμόνιο είναι ένα επίμαχο ζήτημα και θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε κατά πόσον θα πρέπει να παραμείνει στην αδειοδότηση ή στην καταχώρηση. Η Κομισιόν προτείνει, προτεινει πρόκειται να κάνει μια νέα πρόταση και εν ώψη των ψηφοφορίων στην Επιτροπή είπα ότι το Κοινοβούλιο θα παραμείνει και θα εμείνει στο ζήτημα της αδειοδότησης. και προτίθεμαι να παρουσιάσω στην Επιτροπή, στην μας ε, μια πρόταση για μεταβατική περίοδο έτσι ώστε οι χώρες που έχουν το σύστημα διαδότηση να συνεχίσουν με αυτό και οι χώρες που έχουν το σύστημα της καταχώρησης να συνεχίσουν και μετά από μερικά χρόνια να γίνει μια αξιολόγηση και η Κομισιόν να υποβάλει τελική πρόταση. Ό,τι φορά την ε, ανάδεση εξουσιών στην Κομισιόν, παραμένω στην Γενική Συμφωνία που είχαμε μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν. Λοιπόν, Πρόεδρε, αυτά οι συνεχίσεις συνεχίζονται, αλλά έχουμε οδηγηθεί σε άλλη έξοδο. Ευχαριστώ σαφέστατα δεν νομίζω ότι είναι και τόσο καλή η κατάσταση, αλλά συμμετέχουν στον τριμερή διάλογο και τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Ίσως η Δανική Προεδρία που έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τριμερή διάλογο θα ήθελε να μας αναφέρει σχετικά η κυρία Αβε Πουμ, όχι Μάρτιν Σίφερ. αν μπορείτε να σε σαφή την θέση της Κομισιόν και ίσως μετά η Ιδανική Προεδρία να μας πει κάτι και κάποιοι συνάδελφοι ενδεχόμενα να συμβάλλουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι. Στηρίζουμε απόλυτα τον άτυπο τριμερή διάλογο ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή και με τον εισηγητή τον κύριο Μίλτερ και με τη Δανέζικη Προεδρία. Η κατάσταση όπως περιγράφηκε ε, είναι ε, ε, ανταποκρίνεται και στη δική μας αξιολόγηση. Ε, όπως και όλοι οι άλλοι, πάντα δηλώναμε την ευελιξία μας. Η θέση της Κομισιόν όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι συνεχίζουμε να μην ε, στηρίζουμε την διπλή, τη διτή προσέγγιση, ε, θέλουμε ε, αδειοδότηση. Όσον αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης, ε, μένουμε στη θέση που προτείναμε. Ωστόσο, ε, είπαμε ότι στο τρίτο mm. θέμα η εξαίρεση του νητρικού αμμονίου μπορεί, ε, στο θέμα αυτό μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι εφόσον επιτευχθεί ε, συμβιβασμός στα δύο πρώτα μέρη. Αλλά πρόκειται για συνολικό πακέτο, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν έχουν συμφωνηθεί όλα. για να διασαφηνίσω ε, το θέμα αδειοδότησης ε, καταχώρησης. Δύο ε, επιλογές υπάρχουν. Σαφώς η προτιμητέα για μας, όπως υπόθηκε, είναι να, να επιδιώξουμε την αδειοδότηση, αλλά να συμφωνήσουμε πάνω σε μια μεταβατική περίοδο τριών με πέντε ετών και κατόπιν ε, όλα τα κράτη-μέλη να ε, κινηθούν προς ε, την αδειοδότηση, ακόμα και τα κράτη-μέλη που αυτή τη στιγμή έχουν σύστημα καταχώρησης σε εθνικό επίπεδο. Σίγουρα αυτή θα ήταν η προτιμητέα λύση, εάν δεν επιτευχθεί απαραίτητη πλειοψηφία. Η δεύτερη επιλογή θα ήταν να επιδιώξουμε διτή προσέγγιση, να έχουμε αδειοδότηση και καταχώρηση από την αρχή, να Υπάρχει πρόβλεψη όμως για αξιολόγηση μετά από 3 με 5 χρόνια. Και ως μέρος της αξιολόγησης αυτής ε, η Κομισιόν να κληθεί να υποβάλει ε, στη συνέχεια προτάσεις ε, με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των δύο συστημάτων. Η λύση αυτή θα έχει το πλεονέκτημα ότι θα οδηγήσει σε πολιτική που να βασίζεται ακόμη περισσότερο σε στοιχεία. Διότι έτσι θα έχουμε αξιολόγηση και των δύο διαδικασιών, ανάλυση τους σε βάθος και έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε ε, επανεκκίνηση όσον αφορά την εναρμόνιση με βάση περισσότερες αξιολογήσεις. Γι' αυτό αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη λύση, εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η πρώτη. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, εξαρτώνται από την πρόοδο που θα σημειωθεί εδώ στο θέμα αυτό, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να επιδείξουμε την απαραίτητη ευελιξία ε, στο συνολικό αυτό πλαίσιο πολιτικής για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σίφερ. Να ακούσουμε τη Δανέζικη Προεδρία του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Γιάννη Μούλτερ που ε, περιέγραψε την ε, κατάσταση των ε, διαπραγματεύσεων μετά τον επίσημο τριμερή διάλογο που πραγματοποιήθηκε υπό την Πολωνική Προεδρία. Ε, επί Δανικής Προεδρίας δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα επίσημος ε, τριμερής ε, διάλογος. Γι' αυτό είναι δύσκολο να σας πω πώς έχει κατάσταση στο Συμβούλιο και η θέση του Συμβουλίου, αλλά μπορώ να σας πω ότι η Δανέζικη Προεδρία είναι διατεθειμένη να εργαστεί με ανοιχτό και επικοδομητικό πνεύμα μαζί με την Κομισιόν και σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο για να επιτευχθεί μια λύση. Την επόμενη εβδομάδα ελπίζουμε ότι θα γίνει ε, ε, σχετική συνάντηση στο Συμβούλιο που θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Και γι' αυτό σήμερα ακούω προσοχή τα όσα ε, λέει η Επιτροπή ώστε να μπορέσω να δώσω αναφορά στο Συμβούλιο για να βρούμε μια λύση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Μίλτερ για την εξαίρετη παρουσίαση αλλά και για τις διαπραγματεύσεις, οι πολλές συνεδριάσεις των σκιωδών που διοργάνωσε διότι συζητήσαμε επί μακρόν του και η θέση του Συμβουλίου που ε, προκλήθηκε αυτές τις τελευταίες, τελευταίους μήνες ε, κατά τη διάρκεια Προεδρίας γνωρίζει πολύ καλά τα περιθώρια ελιγμών που είναι αρκετά περιορισμένα σε φορά την πολιτική μας ομάδα. Ευχαριστούμε κύριε Μιούντερ για την πολύ καλή παρουσίαση και για την ε, υπομονή σας αλλά και για τις ικανότητές σας. Ευχαριστώ κύριε Βίξτρομ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μυρίζει άνοιξη και μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε σήμερα ή μάλλον χθες. Καλή της ε, ο κόσμος ε, αναπνέει καθαρό αέρα και ε, επίσης ε, καθαρίζει τις πισίνες του. Εδώ υπάρχει πρόβλημα όμως με τις ουσίες. Χρειάζεται να εγγυθούμε την ασφάλεια των πολιτών και η χρήση πρόδρομων εκρηκτικών υλών να περιοριστούν αυστηρώς. Και τώρα προκύπτει ζήτημα καθαρισμού των ε, δεξαμενών ε, κολύμβησης. Ευχαριστώ. Μάλλον να πείτε, Δανική Προεδρία, στο Συμβούλιο ότι αυτό το ζήτημα θα πρέπει να λυθεί και θα πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι καθαρισμού. Πολύ ευρωπαϊκή αυτή η δήλωση για την άνοιξη που βέβαια αφορά και εμάς που δεν έχουμε πισίνα, αλλά τέλος πάντων. Ας ακούσουμε τις αντιδράσεις του κύριου Μούλντερ. Τι βλέπετε, κύριος Μούλντερ. Ενδιαφέρουσα βρήκα τη συζήτηση. Να καθησυχάσω τη συνάδελφο, θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύση για τις πισίνες για μία χώρα συγκεκριμένα και ελπίζουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Σίγουρα πρέπει να κάνουν και οι δύο πλευρές υποχωρήσεις. Προς το παρόν όμως νομίζω ότι τις περισσότερες υποχωρήσεις τις έχει κάνει το Κοινοβούλιο και όχι το Συμβούλιο. Βέβαια μπορεί το Συμβούλιο να έχει διαφορετική άποψη, αλλά ελπίζω η συνεδρία του Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα να σημειώσει κάποια πρόοδο για αυτό το θέμα να μπορέσουμε να λύσουμε το ζήτημα γρήγορα. Γιατί έτσι πρέπει. We thank you. We've had the discussion about the state of play after the trial. Ακούσαμε λοιπόν την πρώτη εργασία μετά τι τριμερεί διαπραγματεύσει. Θα συνεχιστεί η συζήτηση. Χρόνο έχουμε μπροστά μα, αλλά τουλάχιστον προ το παρόν μπορούμε να λήξουμε τη συνεδρίαση και θα επαναλάβουμε τι εργασίε μα στι 3 το μεσημέρι, όπου θα εξετάσουμε τα επόμενα σημεία τη μέσης διάταξη. Γεια σα.